Colleagues, can I bring the meeting to... Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχετε μπροστά σας λογικά την πρόταση για την ημερήσια διάταξη σήμερα και αύριο. Αν είστε ικανοποιημένοι με την πρόταση αυτή, περνάμε στο θέμα το επόμενο, στην έγκριση των πρακτικών πρακτικά της 22ης και 23ης Μαρτίου. Τα εγκρίνετε. Ανακοινώνονται νέες κοινέ θέσεις στις 25 Μαρτίου, στην Ολομέλεια δηλαδή του Μαρτίου, πέρασε η κοινή θέση για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στον τομέα των οδικών μεταφορών, μεταφορών με λεωφορεία και θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα με τους κανόνες, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, οφείλω να σας ενημερώσω για τις νέες αυτές κοινέ θέσεις, κάτι το οποίο μόλις έκανα τα μέλη θα ενθυμούνται ότι είχαμε ζητήσει από τον κύριο Κανσιάν και την κυρία Γιάλα Σέντερ την εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ισπανική Προεδρία επί τη βάση της ψηφοφορίας στην πρώτη ανάγνωση και να θεωρήσουμε τις δύο ψήφους αυτές πακέτο. Έχουν προχωρήσει οι επαφές με την Ισπανική Προεδρία και η συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Το επόμενο θέμα Κοινωνικοί κανόνες στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ράνερ. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Έλα, έχεις το λόγο. Herr Liebe Kollegen, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν τους συναδέλφους ε, για τις ε, επικοδομικές ε, συμβολές τους. «76 συνολικά τροπολογίες είχαμε σε σχέση με αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Άρα λοιπόν εδώ αυτή η έκθεση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και όλο αυτό το θεματικό πεδίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Προσπαθήσαμε εδώ να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα ε, το οποίο δεν θα είναι πολύ δύσκολο αν θέλετε. Οπότε έχω προετοιμάσει τρεις συμβιβασμούς και εκ των προτέρων ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι συμφωνούν με, αυτούς τι προτάσει αυτές τις προτάσεις Ε, όπως σας είπα έχουμε να κάνουμε τρία σημεία. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τις μέγιστες και τις ελάχιστες κυρώσεις, μετά αυτό ήταν για το 10. Για το 17 μετά, σε ό,τι αφορά την πρόταση ε, των πρασίνων, σε ό,τι αφορά μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τις, ε, για τις οδούς των αυτοκινητόδρομους και το σημείο 21, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης. τώρα, από δική μου πλευρά, υπήρξαν, να πω τα εξή, έξι τροπολογίες κατατέθηκαν σε ό,τι αφορά του ασφαλείς χώρους στάθμεσης, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχει εδώ σαφής ανάγκη για ασφαλή υποδομή η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη διαθεσιμότητά της στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν ε, την, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων υποδομών. Σε ό,τι αφορά την ε, δεύτερη πρόταση, να πω τα εξή. Εδώ είχαμε πολλές διαφορετικές απόψεις, δηλαδή για το σημείο 17 αρκεί κανείς μόνο να δει τον αριθμό των τροπολογιών που κατατέθηκαν για να καταλάβει πόσο διστάμενες είναι οι απόψεις. Η πρόταση τώρα ε, αφορά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τις οδούς. Ε, αλλά αυτή η πρόταση διαγράφηκε μέσω αυτής της συμβαστικής πρότασης. Εκείνο που ζητάμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μία ε, αρχή συντονιστική η οποία θα είναι αρμόδια για τον εναρμονισμό ε, και το συντονισμό των ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε το συμπέρασμα τόσο των συζητήσεων όσο και των μελετών τις οποίες έχουμε κάνει. όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ελέγχους ή με τις διαφόρες ε, κυρώσεις, ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αρχή αρμόδια για αυτόν ε, τον έλεγχο. Άρα λοιπόν η σχετική πρωτοβουλία δεν, δεν λαμβάνει συνέχεια στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό αλλά δεν της δίνεται συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να στοχεύουμε σε κάτι τέτοιο και ως δικηγόρος πραγματικά μπορώ να σας πω ότι χωρίς έλεγχο δεν, δεν λαμβάνει χώρα τίποτα. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και τη σημερινή κατάσταση αν δεν προβλέψουμε τέτοιες, ε, τέτοιους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, αυτή η αρχή ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει για να μας δώσει και οδηγίες ως προς το πώς θα μπορούσε να απλουστευτεί το σύστημα επιβολής κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω ε, τη σύμφωνη γνώμη σας σε ό,τι αφορά αυτήν την πρόταση τη συμβαστική, η οποία δηλαδή προτείνει πλέον όχι τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τις οδούς, αλλά μιας συντονιστικής υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε, Έλα, από τους σοσιαλιστές τώρα, κύριε Σερδού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, εμείς ε, προφανώς ε, συζητήσαμε με την εισηγήτρια ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση η οποία θα είναι και λογική σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ της κατευθύνσεις. Ε, κάποια σχόλια τώρα που θα θέλαμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη συμβαστική πρόταση 2. Αυτή η πρόταση η οποία αφορά ακριβώς τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής για τις οδικές μεταφορές, για τις οδούς, εμείς θεωρούμε πως ένας τέτοιος οργανισμός ε, δεν συγκεντρώνει από τη δική μας ε, πλευρά ούτε απόλυτη συνένεση, ούτε απόλυτη απόρριψη. Εκείνο που για μας είναι σημαντικό είναι η τροπολογία μας υπαριθμών 43 άσχετα του τι θα ψηφίσουμε, να γίνει δεκτή. Γιατί στην ε, τροπολογία 43 αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ζητάμε καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη η οποία θα εξετάζει ε, το τι μπορεί να κάνει αυτή η υπηρεσία και σε τι ε, ε, θα ωφελεί αυτή η υπηρεσία. Αν λοιπόν η μελέτη δώσει το αποτέλεσμα ότι ναι χρειαζόμαστε ε, την δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας, τότε καλώς. Αλλά εάν δεν προτύψει κάτι τέτοιο, τότε δεν είμαστε υποχρεωτικά υπέρ της σύστασης ενός τέτοιου οργανισμού. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συμβαστική πρόταση υπαριθμών 1. Und beim Kompromiss Nummer 3. Σε ό,τι αφορά την συμβαστική πρόταση 3 υπάρχει θα θέλαμε μια διευκρίνηση. Μας ε, υπόθηκε ότι εάν γίνει δεκτή αυτή η συμβαστική τροπολογία 3, ε, τότε καταπίπτουν 71 έως 74, αλλά ε, θεωρούμε πως αναφερόμαστε στην 72 έως 74, όχι στην 71, η οποία αντιστοιχεί ουσιαστικά σε αυτή τη συμβαστική πρόταση υπάρχουν 3. Πάντως και σε αυτό το σημείο μπορούμε να συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια. σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία 61. Σε ό,τι αφορά τις ε, διάβλους ενημέρωσης, αν θέλετε, δηλαδή ενημερωτικά φυλάδια, Ε, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ε, οδικών αξώνων ε, έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη η συγχύτρια σε ό,τι αφορά την σύμφωνη γνώμη της, ενώ σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 63, 62 και 64 διαφωνεί. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ αυτών των τροπολογιών και της παρούσας τροπολογίας 61 του κύριου Κοχ. Κατά τα ε, λοιπά μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις υπόλοιπες προτάσεις της συζήτησης και θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για τις εργασίες της. Thank you. Ε, ναι, η συγκέντριά μα δυστυχώ δεν ήταν σε θέση να βρίσκεται εδώ, οπότε θα ήθελα να πάρω εγώ το λόγο εκ μέρου τη. Καταρχήν να ευχαριστήσω εγκάρδια ε, την συγκέντρια τη ε, πρόταση ψηφίσματο. Το ότι εμεί δεν έχουμε υποβάλει τροπολογίε δείχνει ότι ο κόσμο δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θεωρούμε πω είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση και μπορούμε να συμφωνήσουμε με το σύνολό της σε ό,τι αφορά τώρα τις συμβαστικές προτάσεις. Είμαστε σε θέση να τις ε, υποστηρίξουμε όλες. Τα όσα είπε ο κύριος Σόρτουξ σε ό,τι αφορά τον τροπολογία 43 ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή εμείς η ε, 43 θεωρούσαμε ε, πως αποτελεί μια πιο θετική αν θέλετε αντιμετώπιση αυτής της, του ενδεχομένου της δημιουργίας ενό τέτοιου ευρωπαϊκού οργανισμού οδικών μεταφορών αλλά μας εκπλήσει το γεγονός ότι είπατε ότι δεν είσαστε κατηγορηματικά υπέρ γιατί και εμεί έχουμε αυτή την άποψη, ότι ενδεχομένω δηλαδή να μην είναι απαραίτητη σύσταση ενό τέτοιου οργανισμού οδικών μεταφορών. Άρα θα, θα εξαρτηθεί λοιπόν ε, από αυτή την τοποθέτησή μας και το κατά πώ θα είμαστε υπέρ τη ε, συγκεκριμένη συμβαστική πρόταση, δηλαδή από το τι θα γίνει με το 43. Πάντω, στο σύνολό τη συμφωνούμε με αυτή την πρόταση. Ε, κυρία Λίχτενμπεργκερ, πράσινη. Ναι, ε, σχεδόν ε, είμαι μόνο γερμανική αυτή η συζήτηση, έτσι. Αλλά αυτό καταδεικνύει ότι ακριβώς η κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβολή και ερώσεων είναι ιδιαίτερα οξυμένη στις ε, χώρες της ε, κεντρικής Ευρώπης που βρισκόμαστε δηλαδή στο, ακριβώς ε, στο κέντρο γιατί εκεί βιώνουμε περισσότερο τις επιπτώσεις του συστήματος και της κατάστασης όπως είναι σήμερα. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η τροπολογία 31 Lightfield γιατί έχει λάβει αρνητική τοποθέτηση από την εισηγήτρια. Ε, δηλαδή το να ε, συμμετάσχουν σε ειδικές συζητήσεις για τα μέλη της ε, ATR. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί. Γιατί αν δεν εμπλέξουμε αυτά τα μέλη της ATR μέσα στη συζήτηση, τότε υπάρχουν οι κίνδυνοι κοινωνικού ντάμπινγκ και ούτω καθεξής. κάτι. δική μας άποψη λοιπόν πρόκειται για σημαντική τροπολογία και θα έπρεπε να παραμείνει σε κάθε περίπτωση στο κείμενο. Σε ό,τι αφορά τώρα τι συμβαστικέ τροπολογίες, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά το δύο, ε, η ασφάλεια στι οδικέ μεταφορές θα αυξηθεί εάν τα κράτη-μέλη τελικά επιβάλλουν και βάλουν, εστιάσουν σε παραβιάσεις, σε παράδειγμα, της ανώτατης ε, ε, ταχύτητας ή της κατάχρησης αλκοόλ. Ε, να αντιμετωπίσουν δηλαδή τέτοιου είδους φαινόμενα μέσω των κατάλληλων ελέγχων. Εκεί βρίσκεται το, το κυρίω ζήτημα, όχι στην δημιουργία ή όχι ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα με συζητήσεις με σαφή και πρακτικά βήματα. Στον χώρο των οδικών μεταφορών μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Ε, εφόσον δηλαδή εγώ μπορώ να συνεχίζω να οδηγώ όταν είμαι μεθυσμένος σε ένα κράτος μέλος ε, και ε, έχω ε, τη δυνατότητα να αποφύγω το να μου πάρουν την, το δίπλωμα γιατί μπορώ να προσφύγω κατά μία σχετική απόφαση είναι κάτι το οποίο δεν ωφέλη, δηλαδή ειδικότερα σε ό,τι αφορά εκείνους που κάνουν ε, μεγάλα ταξίδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμβαστική τροπολογία 3. Προφανώ αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα ύπαρξη τέτοιων χώρων στάθμευση, αλλά από την άλλη πλευρά ε, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε εδώ τη βάση ότι χρειάζεται χρηματοδότηση από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι χρηματοδοτούμε τελικά πράγματα τα οποία αν θέλετε δευτερεύοντα και όχι τα βασικά ζητήματα δεν μπορούμε να θέτουμε πλέον ε, τέτοιες λύσεις ε, αντί να θίγουμε τα τα προβλήματα. Υπάρχουν ε, και σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. περιβαλλοντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτούς τους χώρους στάθμισης, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες διαρροές ψυχτικών υγρών και που τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμα κι αν αυτές οι διαρροές γίνονται εκτός κατοικημένων περιοχών, ε, μειώνονται πάρα πολύ οι αξίες των σχετικών οικοπαίδων ε, και υπάρχουν πολλά προβλήματα για τους ε, κατοίκους αυτών των περιοχών, των γύρω περιοχών. Άρα λοιπόν αυτή η πτυχή της δημιουργίας χώρων στάθμευσης θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε, να τη λάβουμε υπόψη μας στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι προβληματική αυτή η αναφορά. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την προφορική τροπολογία Voltman Call, να πω το εξή. Η λήψη βουλώσεων από τα inspection bodies, δηλαδή από τι αρμόδιε αρχέ για τι επιθεωρήσει, είναι κάτι το θετικό, αλλά όταν ε, αναφέρουμε εδώ ε, εκπροσώπους από τους ενδιαφερόμενους φορείς ξέρουμε τι θα συμβεί πάλι. Θα έχουμε από ένα σωρό ε, υπηρεσίες, εκπροσώπους και τελικά δεν θα οδηγηθούμε σε αύξηση της ασφάλειας και σε ε, μείωση των παραβιάσεων αλλά αντίθετα θα προωθηθεί τελικά το να συμβαίνουν, να συνεχίζουν να υπάρχουν παραβάσεις. Δυστυχώ αυτό οφείλω να το ομολογήσουμε βάσει τη δική μου εμπειρία. Thank you, Ευχαριστώ. Συγγνώμη που θα σπάσω την αλυσίδα, αλλά θα συνεχίσω αγγλικά. Θα πρέπει να πω ότι σχετικά με τις αρχικές παρατηρήσεις δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Λίχτεμπεργκ. Και το λέγω αυτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι δηλαδή τα προβλήματα φαίνεται να εντοπίζονται περισσότερο για το θέμα που συζητάμε, για τις χώρες και με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια νομοθετική ρύθμιση η οποία είναι ενός τύπου και θα πρέπει να αρμόζει σε όλους. Ένα νούμερο παπούτσι για όλους. Αυτό είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δημιουργεί πρόβλημα. Στην τελευταία συζήτηση που είχαμε γύρω από το θέμα αυτό είπα αρκετά πράγματα, δεν θα επανέλθω. Θα σχολιάσω λίγο τις τροπολογίες όμως. εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες σχετικά με την πρόταση για μια υπηρεσία οδικών μεταφορών. Φαίνεται και με χαρά το σημειώνω ότι απομακρύνεται η πιθανότητα αυτή. Δεν είναι καθόλου μυστικό το πόσο ε, αντίθετο είμαι με την δημιουργία τέτοιου είδους ε, θα έλεγα υπηρεσιών και νομίζω ότι μια τέτοια ειδική υπηρεσία για τις οδικές μεταφορές θα ήταν απώλεια χρόνου και απώλεια χρημάτων φορολογουμένων. Δεν με εκπλήσουν βέβαια κάποιες άλλες προτάσεις οι οποίες έρχονται εναλλακτικά σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση. Έχουμε αρκετές τροπολογίες οι οποίες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπληρώσει τον ρόλο αυτό και όχι από ε, μια άλλη εξωτερική υπηρεσία ή συντονιστικό όργανο. Και γι' αυτό υποστηρίζω αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι οι οδικές μεταφορές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με τις ασφαλείς θέσεις ε, στάθμευσης, νομίζω ότι οι προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι αδικαιολόγητες. Η γενική άποψη είναι ότι η αύξηση της εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων οι κλοπές αυτοκινήτων ή οι κλοπές από το εσωτερικό αυτοκινήτων είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται συνεχώς και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά είναι καλοδεχούμενο. Να μου επιτρέψετε να πω ότι σχετικά με τη δική μου τροπολογία την 75 ενθυμίστε ότι είχε υπάρξει ένα γλωσσικό θέμα και γι' αυτό είχα καταθέσει την τροπολογία αυτή, έτσι ώστε να μιλάμε για την ασφάλεια, την ασφάλεια από την εγκληματικότητα και όχι την ασφάλεια για άλλους λόγους υγιεινής ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια προβλήματα στη μετάφραση αγγλικά προς γαλλικά και τούμπαλιν. Είναι μια απλή διευκρίνηση, λοιπόν, για το τι πραγματικά θέλουμε να ισχύει σε αυτούς τους φυλασσομένους χώρους στάθμευσης. Σχετικά με την επιβολή των κανόνων αυτών, δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερβολικοί και να αποδίδουμε, να προσδίδουμε μάλλον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερη δουλειά από αυτήν την οποία μπορεί να φέρει πέρας. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα για βελτίωση της κατάστασης μέσω των υπηρεσιών της Κομισιόν, αλλά είναι κυρίαρχος ο ρόλος των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και να τα αναλάβουν. Και να μου επιτρέψετε και να θέσω και ένα ερώτημα. Ε, μου έκανε εντύπωση, χαμογέλασα θα έλεγα, στην τροπολογία 1, να υπάρχει μια φράση σε παρένθεση η οποία λέει να λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικοί παράγοντες ή τα, το ΑΕΠ σε σχέση με τις ποινικέ κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν. Νομίζω ότι είναι λίγο αστεία η αναφορά σε γεωγραφικούς παράγοντες. Ας επανέλθουμε στο γερμανικό τρενάκι. Θα σας διαψεύσω με χαρά. Ως εκ τούτου θα μιλήσω γαλλικά. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο ε, για την εξαιρετική της παρουσίαση. Πρόκειται για μια πράγματι πολύ χρήσιμη παρουσίαση και αναζήτησε τις συμβιβαστικές προτάσεις σχετικά με την οδική υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, και όταν είχε γίνει μια σχετική συζήτηση είχε προταθεί να κάνουμε μια πιο εμβαθυμένη συζήτηση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ε, και τις οργανισμούς μεταφορών σε διάφορους τομείς. Ε, και η δική μου άποψη πολύ σύντομα είναι εάν ε, μια, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός υπάρχει μόνο για να εκπονεί έγγραφα και να προβαίνει σε δημοφιλεύσει, δεν χρειαζόμαστε ένα οργανισμό. Εάν όμω ένα τέτοιο οργανισμό μπορεί να αναλάβει συντονιστική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση, γιατί δεν ξέρουμε αν πάντοτε υπάρχει όπως διαπιστώσαμε κάποια τότε ε, θα μπορούσε ε, να έχει κάποια σκοπιμότητα η δημιουργία ευρωπαϊκών οργανισμών. Αλλά αυτό θα σήμαινε ε, μια πολύ εκτεταμένη, πολύ εις βάθος συζήτηση και σε αυτή την Επιτροπή για το συγκεκριμένο ζήτημα αυτών των οργανισμών. Ίσως καλό θα ήταν λοιπόν προς το παρόν να αναφερόμαστε σε μια τέτοια συντονιστική αρχή και όχι σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δικών ε, Μεταφορών ε, και ε, με τον Φίλιπ Μπράτμπορν είχαμε αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου σε εβδομαδιαία επίπεδα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή υπάρχει η κίνηση η οποία έρχεται από διάφορες περιοχές, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και ούτω καθεξής και βλέπουμε ε, πόσο διαφορετικές ε, και με πόση φαντασία δίνονται οι ερμηνείες στις διάφορες ε, διατάξεις. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός εάν θέλουμε να υπάρχουν διαφοροποίησεις. Όταν είχαμε εκπονήσει τη σχετική οδηγία σε ό,τι αφορά το δίπλωμα είχε γίνει μια σχετική συζήτηση. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος όπως η Γερμανία που προβλέπει την, το να λαμβάνεται οριστικά να μην μπορεί να, οριστικά πλέον να χρησιμοποιήσει κάποιος το δίπλωμα οδήγησης. Ε, και μιλάμε για περίπτωση οριστικής Ε, και σε αυτή την περίπτωση της αφαίρεσης ε, του διπλώματος ε, δεν μιλάμε για μια παροδική κατάσταση, είναι οριστική και αυτό ισχύει παντού και δεν ισχύει ό,τι ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη όπου για παράδειγμα η αφαίρεση αυτή ισχύει μόνο για 14 ημέρες και μετά λαμβάνει κανείς το δίπλωμα. Θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να υποστηρίξουμε την πρόταση της συναδέλφου. Ευχαριστούμε κύριο Σαλκαντροή. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Την προηγούμενη φορά είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έπρεπε κάτι να κάνουμε για την ερμηνεία της νομοθεσίας ε, σε αυτό το τομέα. Η τροπολογία 19 λοιπόν της Βορτμαν Κόλ νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική γιατί ζητάει πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με μια διατύπωση ενιαίας και δεσμευτικής ερμηνείας του κανονισμού σχετικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης. Είναι πολύ βασικό αυτό να το επαναλάβουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι καλά διατυπωμένες. Μερικές φορές θα θέλαμε να τονίζουν περισσότερο την ουσία. Πάντως για την τροπολογία 2, όσον αφορά τον οργανισμό ήταν ένα πρώτο βήμα ή θα μπορούσε να ήταν ένα πρώτο βήμα. Θα ήθελα να ψηφίσουμε για τη 43. Πιστεύω ότι κάλλιστα μπορούμε να την ψηφίσουμε γιατί είναι συμπληρωματική. Όπου ζητάω, τη δικιά μου τροπολογία και ζητάω να εκπονήσει μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συγκρότηση ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δικών Μεταφορών. Δεν λέμε αν είμαστε υπέρ ή κατά, λέμε να εκπονηθεί μελέτη για να γίνει συζήτηση, για να αποφασίσουμε τελικά αν τον θέλουμε ή όχι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, το τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω είναι η τροπολογία μου 68, όπου ζητάω να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ώστε οι οδηγοί να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνονται για ό,τι κανόνες οι κυρώσεις επιπαραβάσεων υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Όσο γίνεται περισσότερο λοιπόν να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, όχι μόνο ένα έντυπο, ένα φυλάδιο, αλλά και σε πραγματικό χρόνο να μπορούν οι οδηγοί να ενημερώνονται όσον αφορά τα διάφορα δεδομένα που αφορούν το επαγγελμά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να, να την υποστήριξη μου απέναντι στην κυρία Άραν, ε, γιατί ε, εκπώνησε ε, με εκθέση υψηλή ποιότητα και θα συμφωνήσω με τα όσα είπε ο συνάδελφο κ. Ματιό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού οργανισμού. Είμαι απογοητευμένο που δεν έλαβε την υποστήριξη των συναδέλφων η σύσταση ενό τέτοιου οργανισμού γιατί όπω μόλι τώρα είπε ο συνάδελφο Γκρό έχει νόημα. Έχει νόημα η δημιουργία ενό τέτοιου οργανισμού, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ε, τηρησή των ε, κοινωνικών διατάξεων, ή, ε, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτού του Eurovignette, σε ό,τι αφορά την μείωση της κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά Σαββατοκύριακο και ούτω καθεξής. Θα είχε νόημα η σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού. Εγώ πάντως μπορώ να συμφωνήσω και με τη συμβαστική ε, τροπολογία και με την τροπολογία που αναφέρθηκε από τους συναδέλφους σε ό,τι αφορά την εκπόνηση μιας σχετική μελέτης για τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση, σε ό,τι αφορά τους ε, χώρους στάθμισης, ε, θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν ε, ε, Συμβάλλουμε δηλαδή σωστά ε, σε ό,τι αφορά την καλύτερη κυκλοφορία. Δηλαδή χρειαζόμαστε και για συνθήκες υγιεινής αλλά και για λόγους εξεκούρασης των οδηγών να έχουμε τους απαραίτητους αυτούς χώρους στάθμευσης. Και ε, προφανώ ε, σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση υπάρχουν και ζημιέ οι οποίε ε, προκύπτουν και τι οποίε καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον, την εισηγήτρια, αλλά και τους σκιώδες εισηγητές. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες. Την τροπολογία 57 πρώτα απ' όλα. Πάνω στην οποία θα κάνω μια προφορική τροποποίηση για να διατηρηθεί στο κείμενο μόνο το πρώτο τμήμα όπου λέει ότι η ακινητοποίηση του οχήματο είναι ένα μέτρο έσχατης ανάγκης. Και αυτό για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα γίνονται καταχρήσεις στα διάφορα κράτη-μέλη για να μην υπάρχουν ε, φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, για παράδειγμα. Γι' αυτό το υπόλοιπο, μετά από αυτό που σας ε, ανέφερα, θα το διαγράψω στην προφορική μου τροποποίηση. Και έτσι ελπίζω να με στηρίξουν οι συνάδελφοι. Μια άλλη τροπολογία τώρα. 76. Εδώ Μιλάμε για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων για την κατασκευή ασφαλών χώρων στάθμευσης. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιοι ασφαλείς χώροι στάθμευσης και αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αν θέλουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε την καλή τήρηση των κοινωνικών κανόνων, τότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη ώστε εκείνα να οικοδομήσουν τέτοιους χώρους στάθμευσης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η τροπολογία 76 είναι σημαντική. Έχουμε πειραματικά προγράμματα που τα έχουμε στηρίξει εδώ στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε συνεπείς με την ιδέα αυτή και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο ε, προς αυτή την κατεύθυνση, για την κατασκευή δηλαδή ασφαλών χώρων στάθμευσης. Ευχαριστούμε κύριε Τικάου. Ο κύριος Πασκορέλη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ να μου δώσετε και την ευκαιρία να συνεισφέρω στην γλωσσική ποικιλία στη συνεδρίασή σας ομιλώντας την Ιταλική γλώσσα. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί θετική την ε, έκθεση την οποία εξετάζουμε. Η ανακοίνωση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία βασίζεται η έκθεση υπογραμμίζει αν θέλετε το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στη μία από τους ουσιαστικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και νόμους για τη διάρκεια οδήγησης και ανάπαυσης κτλ. Και από την άλλη με το ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό δεν υπάρχουν τα μέσα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων αυτών γιατί οι αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στα κράτη-μέλη που είναι αποκλειστικοί νομοθέτες ουσιαστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το αφισβητεί αυτό σε καμία περίπτωση, απλά το σημειώνει και ανησυχεί για την κατάσταση, γιατί από πλευρά των κρατών μελών ε, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή εφαρμογή των κανόνων αυτών και να επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες να είναι ανάλογες του προβλήματος. Αυτό το οποίο όμως δυστυχώς διαπιστώνουμε είναι ότι το επίπεδο των κυρώσεων ποικίλει από τη μία χώρα στην άλλη. Οι παραβάσεις ε, κρίνονται διαφορετικά αν είναι σοβαρές ή όχι ανάλογα με το κράτος μέλος και αυτό το δείχνει η έκθεση. Αυτό όμως δεν είναι κριτική ε, την οποία θα πρέπει να στρέψετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση ήταν αυτή εξ αρχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη. Θα πρέπει λοιπόν με τον ε, πιο εναρμονισμένο τρόπο να εφαρμόσουμε τις ρυθμίσεις αυτές χωρίς να παραβιάσουμε τις αρμοδιότητες τις οποίες κατά αποκλειστικότητα έχουν οι χώρες. Σας είπα ότι αυτή είναι η άποψη του νομοθέτη, δεν το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε είναι να κατευθύνουμε τα κράτη-μέλη σε μια κοινή ανάγνωση του κανονισμού, σε μια κοινή αξιολόγηση της βαρύτητας των παραβάσεων και παραβιάσεων και του τύπου των κυρώσεων Εφόσον δεν αλλάζει η νομική ρύθμιση και εφόσον οι κοινέ αρμοδιότητες ή μάλλον η κατανομή των κοινών αρμοδιοτήτων μένει ως έχει, δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σημειώνει αυτό η έκθεση έτσι ώστε να πετύχουμε ε, μια όσο περισσότερο εναρμονισμένη ερμηνεία θα έλεγα των συνθήκων. Η συνθήκη της Λισαβόνας δίδει ορισμένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο συνεργασίας και όχι εναρμόνισης. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά τα πράγματα ως έχουν είναι αυτά τα οποία περιγράφει και η συγγήτριά σας. Δεν θα σχολιάσω τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γιατί πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής σας. Υπάρχουν όμως τέσσερα συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, για την εξωτερική υπηρεσία. Ανεξαρτήτως των θετικών ή αρνητικών χαρακτηριστικών που έχουν οι υπάρχουσες υπηρεσίες, θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ξεκινήσει έναν διοργανικό διάλογο ο οποίος έχει σαν στόχο την αξιολόγηση των υπαρχουσών εξωτερικών υπηρεσιών όπως επίσης και το επίκαιρο ήμι ανάπτυξης νέου τύπου ή νέων γενικότερα εξωτερικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σε μια πρώτη φάση να παγώσει θα έλεγα το θέμα της δημιουργίας των νέων εξωτερικών υπηρεσιών. Το θέμα των χώρων στάθμευσης είναι ένα θέμα το οποίο ε, πράγματι ε, βιώνουν με δύσκολο τρόπο οι επαγγελματίες, οδηγεί Γνωρίζετε επίσης ότι μετά και από δική σας πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει κάποια προγράμματα πιλωτικά για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας, ε, την security δηλαδή και όχι τη safety όπως είπε πολύ σωστά ο Bradborn Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια γενικότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από το θέμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά οι πιστώσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το ε, περιφερειακό ταμείο, όπως επίσης ε, και οι δημοσιονομικές πιστώσεις για τα δίκτυα αυτά, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εν μέρη και για την ενίσχυση αυτού του πακέτου σχετικά με την τροπολογία 31, Lightfried, για το ATR, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε. Πράγματι η τροπολογία αυτή έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Γιατί, όπως ε, έχει ήδη ζητηθεί από το Συμβούλιο στο παρελθόν όταν έγινε δεκτός ο κανονισμός για τις ώρες οδήγησης, ώρες ανάπαυσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε στη Γενέβη με όλα τα μέλη του ΠΟΕ την ευθυγράμμιση με τον δικό μας κανονισμό. Έχει ήδη ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τον πρόεδρο κύριο Κώστα και νομίζει ότι έχει κάνει αυτό το οποίο ε, θα έλεγα έπρεπε να κάνει και οι διεθνείς ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις είναι απόλυτα συμβατές και παραλληλίζονται πλέον με τις κοινοτικές ρυθμίσεις. Τέλος, η κυρία Λίχτεμπεργκερ αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά θέματα της οδικής ασφάλειας που αφορούν τα ποσοστά του ινοπνεύματος κτλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα όργανα τα οποία επιβάλλουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να το πετύχουν. Αυτές οι πλευρές της οδικής ασφάλειας θα πρέπει ε, δεόντως να λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση νέων νομοθετικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, δόκτωρα Πασκουαρέλη. Ράνερ θα πρέπει να απαντήσει. Έχουν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι συμπληρωματικέ ερωτήσει. Ε, πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν πολύ σύντομα, όχι με τη σειρά με την οποία τέθηκαν, αλλά με τη σειρά που σημείωσα αυτά τα ερωτήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη μελέτη για τη σκοπιμότητα του οργανισμού και τον οργανισμό γενικά, μου είπαν πως ενδεχομένως αυτό το σημείο εδώ, αυτή η έκθεση δεν είναι το ενδεδειγμένο σημείο στο οποίο θα έπρεπε να κάνουμε αυτέ τι συστάσει ε, περί δημιουργία ενό τέτοιου οργανισμού. Αυτό μπορεί να γίνει κάπου αλλού. Θα μπορούσαμε έτσι ω αρχή να αναφερόμαστε σε αυτήν την ε, συντονιστική υπηρεσία. Ίσως θα πηγαίναμε πολύ μακριά εάν κάναμε ήδη λόγο για ευρωπαϊκό οργανισμό. Μπορούμε να κάνουμε λόγο ε, για μια συντονιστική αρχή και αργότερα να μεταβούμε στην πρόταση για έναν οργανισμό. Υπό Αυτές τις συνθήκες όμως και αφού συμφωνούμε σε ό,τι αφορά το ελάχιστο, ναι, η μελέτη η οποία κοστίζει και κάποια χρήματα θα μπορούσε να εκπονηθεί μέσα στο, μέσα στο μέλλον. Αλλά επειδή σας λέω ε, χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εκπονηθεί ε, και είναι υψηλό το κόστο ε, και η προστιθέμενη αξία μπορεί να μην ήταν μεγάλη, θα μπορούσαμε να μην έχουμε την ακόμη μα τέτοια μελέτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την 43 ήδη έχει περιληφθεί στην Συμβαστική Τροπολογία 3. περιλαμβάνει δηλαδή και την 71 η οποία καταπληκτική αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία 61, πρόκειται για μια επιπρόσθετη τροπολογία, η οποία ε, αναφέρεται στο 20α. Εγώ θα ήθελα, ε, πέραν δηλαδή των τεχνικών δυνατοτήτων, ε, να έχουμε ένα φυλάδιο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, άλλα μέσα, τεχνικά μέσα βοήθειας, ούτως ώστε σε σχέση και με την τροπολογία 68 να καθίσταται σαφές γιατί θέλουμε να γίνεται μια τέτοια αναφορά. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 31 του συναδέλφου Λάιφριντ, μου είπαν πως έχει αποσυρθεί. Μας το είπε δηλαδή. ο ε, Λάιφριντ για τους λόγους που ανέφερε και ο συνάδελφος. Ε, πραγματικά νομίζω πως εργαζόμαστε παράλληλα και δεν με χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος το είπε άλλωστε, ο συντάκτης δηλαδή της τροπολογίας, ότι την αποσύρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους χώρους ε, στάθμες, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δηλαδή ε, ε, δεν... Ε, σημαίνει ότι εάν δεν έχουμε χώρους στάθμευσης μπορούμε να προωθήσουμε άμεσα με άλλους ε, τρόπους ε, τις οδικές μεταφορές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι χώροι στάθμευσης οι οποίοι θα πρέπει να προστατευτούν και από εκεί και μετά προφανώς και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την επέκταση των συνδρομικών μεταφορών, ειδικά μετά από τα όσα είδαμε και με το πρόβλημα με το ηφαίστειο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τις ε, χώρες της υπηρετικής Ευρώπης, τα, οι οποίες θεωρούνται ως ε, χώρες διάλευσης, πράγματι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα, λοιπόν, ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τέτοιου είδους παράγοντες μέσα στο σύστημα επιβολής κυρώσεών τους και να μπορούν να προβαίνουν σε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε συνάδελφος Ετικάου και το μπλοκάρισμα των ε, φορτηγών. Προφανώ αυτό ε, θα μπορεί να είναι μόνο το αυστηρότερο μέτρο που μπορεί να επιβληθεί. Αυτό δηλαδή είναι, είναι, είναι σαφέ. δηλαδή σε ό,τι αφορά το σύστημα κυρώσεων το οποίο πρόσφατα μα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν δηλαδή και διάφορε κλίμακε διαφορετικέ. Εκείνο το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω και το οποίο μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα είναι μέτρα εναρμόνιση και ε, διευκόλυνση τη εναρμόνιση αυτών των μέτρων μέσω κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη-μέλη. Τώρα, όταν λέει ο κ. Πασχαλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει το πρόβλημα ε, σε σχέση με τις εθνικές διατάξεις. Προφανώς και το γνωρίζω αυτό σε δικηγόρος ειδικά, ε, το πόσο δηλαδή δύσκολο είναι να ε, παρέμβει κανείς στις εθνικές διατάξεις των κρατομελών. Αυτό όμως που κάνουμε εμείς εδώ είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες δυνατότητες εδώ για μέτρα τα οποία επιφέρουν εναρμόνιση και εν πάση περιπτώσει μειώνουν μερικώς τις ε, διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα. Νομίζω πω μερικώς εν μέρη μπορεί αυτό να επιτύχει. Προφανώ, ε, με πραγματήρια ε, δεν πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε έναν κοινό ε, παντελώς εναρμονισμένο κατάλογο κυρώσεων. Και προφανώ είναι και λογικό ότι με βάση τα διαφορετικέ ανάγκε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τι δικέ του κυρώσει, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και ένα ανώτατο όριο, αν θέλετε. Το ίδιο ισχύει ε, ή μάλλον αυτό απηχείται ακόμα καλύτερα με τη συμβαστική πρόταση 1, δηλαδή την επιβολή ελάχιστων και μέγιστων ε, κυρώσεων. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για τι προτάσει σα μέσω των συμβαστικών τροπολογιών ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ε, ίδρυση του οργανισμού και τη μελέτη, έχουμε προβεί σε ανταλλαγή απόψεων. Απλώς σας λέω, δεν ε, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να ε, αναφερόμαστε στην εκπόνηση της ε, μελέτης εδώ, χωρίς να λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι απαραίτητη. Εάν βούμε πιο συγκεκριμένα στο, στην εξέταση του ενδεχομένου για την ίδρυση ενός οργανισμού, θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε μια αναφορά στην εκπόνηση σχετικής μελέτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα, έξι μου είπαν ότι θέλουν να επανέλθουν, να πάρουν το λόγο για να ρωτήσουν την κυρία Ράνερ ή για να ρωτήσουν κάτι τον κύριο Πασκαρέλη. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι πριν ζητήσει το λόγο ο κύριος Πασκαρέλη, κανένας δεν είχε ζητήσει το λόγο. Τώρα έξι έχουν ζητήσει το λόγο αφού ακούσαμε τον κύριο Πασκαρέλη. Εντάξει. Ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Μπράντμπορ όμως προηγουμένως έχει διαδικαστικό εκτός αν δεν είναι ακριβώς διαδικαστικό. Ναι, ναι. Η κυρία Ρανέρ δεν αναφέρθηκε στην απάντησή της καθόλου στο θέμα της ασφάλειας ε, από εξωτερικούς παράγοντες ή της ασφάλειας που έχουν να κάνουν με αυτό καθε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να γίνει μια γλωσσική διευκρίνηση εδώ. Ναι, ναι. Γνέφει καταφατικά ότι θα είναι security. Με τη σειρά. Ένα λεπτό καθένας. Μάισνερ πρώτα. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Απλά ε, ξέχασα να αναφέρω κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρει η πολιτική μου ομάδα σε ό,τι αφορά την πρωτοπολογία ε, 68 του Αλχαντρού. Ναι, θεωρούμε θετικά η οδηγή των φορτηγών να ενημερώνονται στα σύνορα σε σχέση με τα όσα ε, μπορούν να ισχύουν, αλλά αυτή η αναφορά που γίνεται στα συστήματα προσδιορισμού θέση GPS δεν είναι απαραίτητη. Αυτό ε, ξέχασα να αναφέρω στην προηγούμενη παρέμβαση. Ευχαριστούμε κυρία Λίχτεμπεργκερ. μία μόνο παρατήρηση θα κάνω ε, Κύριε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και εκείνης διαδικασιών ε, κατά παράβαση σε περίπτωση που υποψιάζεται ότι υπάρχει μια τέτοια παράβαση και αύριο θα γίνει και μια σχετική συζήτηση καθώς ε, η συνέπεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν εδώ εκκλήσεις, υπάρχουν αξιώσεις απέναντι στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. συνέπειες. Ε, και να σας πω κάτι, εμείς στην Αυστρία λαμβάναμε πάντοτε διαδικασίες τέτοιες όταν προβαίναμε σε έλεγχο, όχι όταν δεν προβαίναμε. Ε, Ο κύριος θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι σχετικά με τον οργανισμό μου που προτείνω. Πρώτα απ' όλα. Δεν ήταν δικιά μου ιδέα η πρόταση αυτή. Η ίδια η εισηγήτρια στην αρχική της έκθεση και ο συντονιστής του ΕΛΚ στη δικιά του έκθεση το προτείνανε. Εγώ προσπάθησα να κάνω ένα συμβιβασμό και να ζητήσω μια μελέτη για αυτόν τον οργανισμό. Και κάτι ακόμα. Η δικιά μου τροπολογία 43 δεν καταπίπτει άμα ψηφίσουμε το συμβιβασμό, παραμένει δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσει η συγκίτρια. Η συγκίτρια μπορεί να πει ότι συμφωνεί, δεν συμφωνεί με αυτή την τροπολογία. Είναι ελεύθερη να μην την υποστηρίξει. Αλλά αυτό που εγώ υποστηρίζω είναι ότι δεν καταπίπτει και ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους συναδέλφους να ψηφίσουν πάνω σε αυτή την τροπολογία. Το λέω αυτό ρητά στη γραμματεία, να το έχει υπόψη της, ότι η τροπολογία 43 πρέπει να τεθεί στην ψηφοφορία και μετά θα δούμε κατά πόσο θα περάσει όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στέρτοκ. Υποστηρίζω ε, τα όσα είχε αναφέρει ο Σάρβο ο σε στη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά θα ήθελα να ε, σα εμπιστεύσω την προσοχή σε μια λεπτομέρεια εδώ, γιατί ε, μπερδεύτηκα εδώ λίγο σε ό,τι αφορά τη χρήση του όρου στη δονηστική αρχή. Στην τροπολογία 55 έχουμε μια ερετική τροπολογία του συναδέλφου Κοχ, που θέλει να αντικαταστήσει τη χρήση του όρου ε, συντονιστική αρχή με τον όρο επιτροπή. Τελικά σε τι θα κάνουμε αναφορά, σε συντονιστική αρχή ή σε επιτροπή, για να ξέρουμε δηλαδή πάνω σε ποια βάση θα συνεχίσουμε να συζητούμε αυτό το ζήτημα. Finally, Mr. Καλώς, τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα μιλήσω πολωνικά ακριβώς για να συνεχιστεί η ποικιλομορφία η γλωσσική εδώ. Το θέμα των θέσεων στάθμευσης είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά προσοχή, μην φτιάξουμε ειδικό οργανισμό γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι έτσι πολλαπλασιάζουμε τους οργανισμούς που ήδη υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι θα πούν οι Ευρώσκεπτικιστέ, ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσθέτουμε επιτροπές, υπηρεσίε, οργανισμούς. Εγώ ξέρω την κυρία Ράνερ και πιστεύω ότι θα είναι λογική και θα καθίσει και θα υπολογίσει το κέρδος και το κόστος. Μην ξεχνάμε ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος θα πληρώνει όλα αυτά. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, κυρία Ράνερ, αν θέλει να απαντήσει για το θέμα του κατά πόσο πρόκειται για μια συντονιστική υπηρεσία για την Επιτροπή ή για μια Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι θα φτιάξουμε οργανισμό για ασφαλή θέση στάθμευσης. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Κύριε Ράνερ. Στη συμβαστική πρόταση γινόταν αρχικά λόγος για ένα εργαλείο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά στην ε, Τροπολογία Κοχ. Das wird mit einem oral Γίνεται τροποποίηση με ρητή τροπολογία και θα πρέπει απλά να γίνει αλλαγή σε επιτροπή. Του όρου επιτροπή. Δηλαδή, αν διαβάσει κανεί την ε, τροπολογία 55, διαπιστώνει κανείς αυτή την ε, αλλαγή. Προφορική λοιπόν ε, τροπολογία σε ό,τι αφορά αυτή την τροπολογία 55 για την αλλαγή αυτού του όρου σε επιτροπή. Δηλαδή λέτε ότι με την προφορική τροπολογία γίνεται επιτροπή όρος αντί για αυτόν που έχουμε εδώ. Ωραία, Οι περισσότεροι μπορεί να είναι κατά της προφορικής ε, τροπολογίας, οπότε έτσι να ψηφίσουμε την αρχική γραπτή τροπολογία. Ωραία. Δεν ξέρω αν κανείς είναι κατά της Επιτροπής ο σώμα. Αν μη τι άλλο δύο εδώ μέσα θα έχουν διαφορετική άποψη. Τέλος πάντων, κύριε Πασκαρέλη, έχετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, ωραία, ευχαριστώ γιατί ειλικρινά δεν θα ήθελα να έχουμε άλλου έξι που ζητάνε το λόγο μετά από εσά. Δεν λέω ότι εσεί φταίτε, δεν λέω ότι είναι δικό σα λάθο, όχι. Αλλά Βλέπετε οι παρεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουν και τους βουλευτές εδώ να θέλουν να πούνε κάτι μετά. Σας ευχαριστούμε. Πάντως, ευχαριστούμε την κυρία Ράνερ. Αύριο ψηφίζουμε την έκθεσή σα. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα είναι τα πρότυπα για τις επιδόσεις των καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο κύριος Φλάσακα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Παρακαλώ, εφόσον θέλετε να βγείτε όσοι βγείτε, να προσπαθήσετε να το κάνετε με κάποια ησυχία. Συγγνώμη κύριε Βλάσσακ. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική. Ήδη από το 1995 υπήρξε μια σαφή στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και το 2007 υπήρξε μια εντελώ διαφορετική νέα απόφαση για τη μείωση των καυσαερίων 20% μέχρι το 2020. Οι προσπάθειες τις οποίες κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσονται στην συγκεκριμένη αυτή τάση μείωσης της εκπομπής καυσαερίων. Και αυτό ισχύει και με τις προτάσεις στον τομέα των LCV, δηλαδή των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων, οχημάτων. Το θέμα το οποίο συζητάμε επηρεάζει σαφέστατα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του αέρα που αναπνέουμε, όπως επίσης και τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσης. Όπως επίσης και κάνει προτάσεις για την αύξηση ε, του αριθμού των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Γι' αυτό λοιπόν οι στόχοι τους οποίους θέτει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεσοπρόθεσμη μείωση των ρήπων που εκπέμπουν τα μεσαία ή ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είναι θετικές οι προτάσεις αυτές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά πράγματα και χάρη στην δική μας πίεση, την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει υπάρξει μια ουσιαστική μείωση ε, των εκπομπών ακόμα και πριν από την επιβολή θα έλεγα απόλυτα δεσμευτικών προτάσεων για τα μέτρα μείωσης. Από την άλλη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσπάθεια την οποία κάνουμε δεν θα πρέπει να είναι μια μονομερής προσπάθεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα. Στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και αναφέρομαι στο 15 με 16% των οχημάτων που κυκλοφορούν γενικότερα, ο κύκλος ζωής των οχημάτων αυτών δεν ξεπερνά τα 10 χρόνια. Μετά από τα 10 χρόνια υπάρχει ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις ε, της ε, ε, σοβούσης οικονομικής κρίσης, τα ανεπαρκή έσοδα των επιχειρήσεων, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανανεώσεις των στόλων αλλά και την έρευνα και για την ανάπτυξη που απαιτείται στον τομέα αυτό. Αυτό έχει μικρότερη χρήση των οχημάτων, έχει οδηγήσει και σε μικρότερη ζήτηση και αύξηση των τιμών των οχημάτων αυτών, τα οποία καθίστανται λιγότερο ελκυστικά για τις ε, επιχειρήσεις ε, οι οποίες τα απασχολούν και για τους χρήστες γενικότερα. Παράλληλα, η πρόταση αυτή βασίζεται και σε συζητήσεις με ερευνητικά κέντρα, με παραγωγούς, με ε, πανεπιστήμια και με τους χρήστες των ε, οχημάτων αυτών. Εγώ είχα οργανώσει μια στρογγύλη τράπεζα στην Τσεχία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων της ε, Ομοσπονδίας Κατασκευαστών τέτοιων οχημάτων αλλά και ερευνητικών κέντρων. Αν σας ενδιαφέρουν οι παρουσιάσεις που έγιναν σε αυτή τη συζήτηση, με πολύ μεγάλη χαρά θα σας δώσω τα πρακτικά. Τι προτείνουμε λοιπόν να συγκεκριμένα από εδώ και πέρα μετά από τις επαφές που είχαμε με την αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. Θέλουμε οι στόχοι να γίνουν ε, ρεαλιστικοί και θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να συνδέονται και με την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων. Οι προτάσεις που κάνουμε είναι οι εξής. Καταρχάς, η θέση σε ισχύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αναβληθεί ε, για μία τριετία σχετικά με τον στόχο των 175 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Ο στόχος για το 2020 θα πρέπει να μειωθεί από 135 γραμμάρια σε 162 γραμμάρια και προτείνουμε επίσης και περαιτέρω μέτρα. Τα έσοδα από την επιδότηση αυτή που από τα χρήματα τα οποία θα προέλθουν από την επιπλέον εκπομπή θα χρηματοδοτήσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εκπομπών. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές ε, ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων. Η κατάσταση έχει ως εξή. Το Συμβούλιο έχει μια μεγάλη ευθύνη τώρα πλέον γύρω από την υπόθεση αυτή. Το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει σε μια συγκεκριμένη απόφαση γιατί ορισμένες χώρες ανησυχούν για το κατά πόσον τα μέτρα αυτά είναι ρεαλιστικά. Γι' αυτό και η Ισπανική Προεδρία δεν θέλει σε αυτή τη φάση να συνεχιστεί η συζήτηση και απλά αναμένει από την θέση, την θέση μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε πιστεύω τώρα την δυνατότητα να βρούμε κάποιες ε, κοινέ απόψεις και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων για ένα τέτοιο θέμα αρκετά περίπλοκο όλο αυτό τον καιρό και καλό θα είναι να προσέξουμε ότι, να τονίσουμε μάλλον ότι οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας και θα ευνοήσουν χώρες όπως η Ιαπωνία να πάρουν μεγαλύτερα τμήματα των αγορών μας. Ευχαριστώ κύριε Βλάσεκ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Κύριε Ζρίκη, ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τη δουλειά του πάνω σε ένα θέμα που είναι πολύ λεπτό. Εδώ διεκδεύονται θέματα και περιβαλλοντικά και οικονομικά. Είναι λεπτό, λέω το θέμα, γιατί θέτει δεσμευτικά όρια, προδιαγραφές και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και όσον αφορά τις κυρώσεις. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να αμφισβητήσει τα νούμερα αυτά που αποτελούν και το πρόβλημα. Κανένας δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στις οδικές μεταφορές, εννοείται. Ξέρουμε ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, γιατί μόνο εκεί εξακολουθούν να αυξάνονται οι εκπομπές και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είναι στο επίκεντρο. Τώρα, από αυτά που απογραμμίζει ο συγητής πρέπει να δούμε τι στόχο έχουμε και πότε θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Όσο στόχο είναι πιο δύσκολος και όσο πιο σύντομη είναι η προθεσμία για να τον πετύχουμε, τόσο περισσότερο πιέζουμε τη βιομηχανία και μερικές φορές δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και όλα και να επιτύχει το στόχο αυτό. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε νέους κινητήρες ναι, και νέες διαδικασίες για τους κινητήρες που ήδη υπάρχουν, αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Έχουν καθοριστεί δύο. Είναι για τα 120 και μετά για τα 135 γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, πρώτα απ' όλα, για να επιτευχθεί το πρώτο νούμερο που είναι ε, ο στόχος του 175 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, χρειάζεται πολύς χρόνος για να προσαρμοστούν οι κινητήρες. Και στη συνέχεια χρειαζόμαστε ένα, μια νέα γενιά κινητήρων για να πετύχουμε τον επόμενο στόχο των 135. Οπότε, ας πούμε όχι σε τρία χρόνια, ας πούμε ας αφήσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά 135 γραμμάρια να το πετύχουμε το 2020. 2020 γιατί, γιατί η ημερομηνία για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τότε ή που πρέπει να πούμε 162 γραμμάρια το 2020 ή αν θέλουμε να επιμείνουμε για τα 135 γραμμάρια, τότε να πούμε δεν θα είναι το 2020 αλλά αργότερα. Οι οικονομικές επιπτώσεις πέφτουν πρώτα απ' όλα στους ώμους των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό οικονομικό τομέα είναι αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξάγει κτλ. Και έπειτα πολλέ φορέ έχουμε μικρέ και μεσαίες ε, επιχειρήσει που χρησιμοποιούν τέτοιου είδου οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ή είναι πυροσβεστικοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι πιέζουμε οικονομικά και την βιομηχανία, αλλά και του χρήστε των οχημάτων αυτών. Σίγουρα θα γίνουν πολλές συζητήσεις και για την προθεσμία και για ε, την ποσότητα γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο. Υπάρχει και κάτι που δεν αναφέρεται στην έκθεση και αυτό είναι η ταχύτητα. Σημαντικό στοιχείο. Τα οχήματα αυτά έχουν ισχυρό κινητήρα γιατί φέρουν φορτίο που πολλές φορές είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με το ίδιο το βάρος του οχήματος. Μερικές φορές βέβαια δεν έχουν καθόλου φορτίο. Οπότε τότε ο κινητήρας μπορεί να έχει επιδόσεις πολύ μεγαλύτερες. Ποια είναι η συνέπεια. Το ένα είναι ότι τίθεται θέμα ασφάλειας και το άλλο είναι ότι τίθεται θέμα ε, ρήπανσης της ε, ατμόσφαιρας γιατί τότε ξεπερνάνε τα όρια. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ΙΧ και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι στις διατάξεις να συμπεριλάβουμε όχι μια κύρωση υποχρέωση αλλά μια τροποποίηση. Να πούμε ότι εάν οι κατασκευαστές έχουν έναν, ε, ένα σύστημα που περιορίζει την ταχύτητα, αυτό να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ε, οχημάτων αυτών. Είναι ένα καυτό ζήτημα. Συνήθως δεν θέλουμε να το φύγουμε, οπότε μπορούμε να πούμε ότι σε θελοντική βάση να μπορεί να γίνει η τροποποίηση αυτή. Βλέπω εδώ το σφυράκι του Προέδρου να ετοιμάζεται να κατέβει. Έπειτα, για τους ε, μικρούς κατασκευαστές, να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες παρεκκλήσεις στην περίπτωσή τους. Έπειτα, όπως είπαμε, αλλάζουν οι επιδόσεις των οχημάτων ανάλογα με την πλατφόρμα που διαθέτει το όχημα και πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά τις κυρώσεις για τα οχήματα αυτά. Και συμφωνώ με τον εισηγητή, δηλαδή τα χρήματα που θα πάρουμε από τα πρόστιμα για τις κυρώσεις να τα χρησιμοποιήσουμε για καλούς σκοπούς, για βελτίωση δηλαδή έργων που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων επί των μεταφορών από τις εκπομπές του Άφρακα. Ευχαριστώ, λεπόμενο μιλήτριο και τον εισηγητή. Και θα ήθελα εδώ να σας πω ότι φυσικά και είναι ένα σημαντικό εγγραφό αυτό που εξετάζουμε και μάλιστα πολύ σημαντικό για τις μελλοντικέ οδικές μεταφορές που αποτελεί και μια από τις κυριότερες, τη δεύτερη βασικά πηγή ε, προβλημάτων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε ιδιαίτερα φιλόδοξοι σήμερα μάλιστα που θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Δεν συμφωνούμε με τον κύριο Φλάσικ για τις, τις ίδιες ανησυχίες. Υπήρχε το 6% το 1999 μέχρι το 2004. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι και γι' αυτό συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μειώσεις εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ούτε και συμφωνώ για την αναβολή των σημαντικών μειώσεων μέσα σε τρία χρόνια. Εγώ καταλαβαίνω βέβαια τις ανησυχίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση. Πρέπει να μείνουμε στο στόχο. γιατί όταν μιλάμε για μείωση διατρία μέχρι το 2020 ουσιαστικά, υπάρχει και τεχνολογία η οποία εξελίσσεται. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. αυτό και Η αυτοκινητοβιομηχανία εξάλλου τους γνωρίζει τους στόχους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση από το 175 το 2012 και 160 Και δεν βλέπω γιατί να αναβάλουμε για τρία χρόνια την ημερομηνία αυτή, όπως προτείνεται στην έκθεση του συγκητή. Ούτε συμφωνούμε με την πρόταση αντί για 135 να είναι 162 γραμμάρια διοξίδιο του άνθρακα ένα χιλιόμετρο το 2020. Γιατί έχουμε και την ρύθμιση για τα επιβατικά οχήματα και τότε θα ήταν σε αντίφαση αυτά τα δύο. Εννοείται ότι πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν σε επαφή μαζί μου διάφοροι κατασκευαστές αυτοκινήτων Εγώ όμως πιστεύω ότι εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ποιος είναι ο ρόλος μας στην ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος και να μείνουμε σε αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι οι κυρώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε 160 ευρώ αυτό το πρόστιμο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι για τις επιχειρήσεις προτιμάνε να πληρώνουν το πρόστιμο αντί να τηρούν ε, τους κανόνες. Ας δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το όριο ταχύτητας. Να πούμε 100 ή 120 την ώρα. Μειώνοντας την ταχύτητα, μειώνονται και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα 108% και βελτιώνεται και ασφάλεια εννοείται και η χορύπανση. Οπότε έχει νόημα να συζητήσουμε και τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους φιλελευθέρους, ο κύριος Τέρξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέρφους. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε εδώ όπως έχουμε κάνει και με τα επιβατικά οχήματα να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Είπε όμως ο συνάδελφος και ότι για το πρώτο στάδιο, το 175, είναι μια βελτίωση σε σχέση με το σημερινό σύστημα. Νομίζω λοιπόν εδώ ότι πρέπει να μείνουμε στην πρόταση που γίνεται. Να είμαστε αυστηροί, ναι. Να έχουμε απαιτήσει από την αυτοκίνητο βιομηχανία. Δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν πράγματα δυσάρεστα για ορισμένους. Θα ακούσουμε διάφορα παράπονα, διάφορες διαμαρτυρίες. Αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, τότε πρέπει να εμείνουμε στα στοιχεία αυτά. Κάτι άλλο για τον επόμενο στόχο του 2020 και τα 135 γραμμάρια, εδώ τίθεται αλλιώ το ζήτημα. Εδώ δεν ζητάμε μια βελτίωση των σημερινών συστημάτων, ζητάμε να έχουμε στη θέση μας κάτι καινούριο. Και μπορεί να καταλαβαίνω πολύ καλά, γιατί και εμένα μου ήρθαν διάφοροι κατασκευαστές και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το επιχείρημα, αλλά οι δυνατότητες που έχουμε ο κύκλος παραγωγής δεν ε, αλλάζει τόσο γρήγορα, δεν προχωράει τόσο γρήγορα. Οπότε πρέπει να δούμε τον συνδυασμό αυτό, 135 γραμμάρια το 2020. Μήπως είναι δύσκολο. Και στην ομάδα μου πρέπει ακόμα να το συζητήσουμε. Σίγουρα στην κάθε ομάδα κυκλοφορούν διαφορετικά νούμερα, αλλά αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Εκεί που δεν συμφωνώ και με δυσκολεύει είναι ο κατασκευαστής, ο οποίος φτιάχνει το αυτοκίνητο, τον, ε, κινητήρα, την εξάτμιση και μετά προσθέτει κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι οι κατασκευαστές και οι χρήστες πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Τα... Οι τώρα, τα πρόστιμα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Και να συ γι' αυτό θέλω να συζητήσω το θέμα της ημερομηνία. Αν υπάρχει μια αυστηρή απέτηση, 135 γραμμάρια δηλαδή, τότε ίσως να ε, συζητήσουμε για την ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να μειώσουμε τις κυρώσεις, γιατί τότε είναι σαν να δίνουμε κίνητρα να γίνονται παραβάσεις. Οπότε δεν συμφωνώ με όλα με τον κύριο Βλάσικ, αλλά παρόλα αυτά θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έκανε. Ευχαριστούμε για τους πράσινους, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω πως ε, θα αποτελέσει έκπληξη το γεγονό ότι εγώ δεν ε, συμφωνώ με αυτές τις προτινόμενες αλλαγές και θα αναφέρω εδώ κάποια στοιχεία. Ε, το ποσοστό στον συνολικό στόλο αυτών των ελαφρών επαγγελματικών ε, θα αυξηθεί γιατί ακριβώς δεν υφίσταται όλες τις υπόλοιπες απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν. Ταυτόχρονα το εμπόριο μέσω του διαδικτύου ε, αναπτύσσεται και αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί περισσότερη κυκλοφορία, περισσότερες μεταφορές, κυρίως οδικές. Και αυτό έχει τις δικές του επιπτώσεις. Τρίτον, δεν θεωρώ Ε, πως εδώ η, η, η, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δηλαδή και την χρήση αυτών των ε, οχημάτων τα πράγματα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι ε, στον χώρο των βαδικών. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δεν εντάσσονται σε κάποιες τυποποιήσεις αλλά τα ελαφρά επαγγελματικά τα οποία κινούνται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από ότι τα επιβατικά σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημιουργία προβλημάτων στη κυκλοφορία, σε ό,τι αφορά τι ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους, ε, την τήρηση ε, ε, χρόνων ξεκούρασης και ούτω καθεξής. Άρα δηλαδή σε ό,τι αφορά την τήρηση των σχετικών κανόνων τα πράγματα είναι χειρότερα από ότι στον χώρο των επιβατικών, όχι ότι καλύτερα. Και ο, ο στόχος μας είναι Ε, ε, ποιος, ότι θέλουμε να έχουμε λιγότερη κυκλοφορία. Αλλά το πρόβλημά μας είναι ακριβώς αυτό, η κυκλοφορία είναι που δημιουργεί ε, περισσότερη ρήπανση. Τώρα μου αποτελεί κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να προωθήσουν περισσότερη κυκλοφορία. Τότε ας πούμε δεν θέλουμε να έχουμε αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ή της ρήπανσης. Ε, δηλαδή, ε, πολύ συχνά η φύση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη από τους ε, συναδέλφους που ακολουθούν αυτή την οδό. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, γιατί θα πρέπει εδώ να δώσουμε το απαραίτητο κινήτρο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μπορούμε να προστατεύσουμε μέχρι τελική πτώση, δηλαδή μέχρι να συμβεί το αντίθετο ε, με την αυτοκινητοβιομηχανία μα, όπω είχαν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή η ανάπτυξη διασφαλίζεται μέσω ε, κινήτρων, μέσω ε, κατευθύνσεων που δίνουμε. Και μία τέτοια κατεύθυνση πρέπει να είναι η μείωση τη ρήπανση. Δεν αντιλαμβάνομαι το γιατί θα πρέπει εμείς τώρα για μία ακόμα φορά να υποχωρήσουμε, ούτω ώστε μία συγκεκριμένη και κατηγορία οχημάτων που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς να έχει τη δυνατότητα να ρηπαίνει ακόμα πιο πολύ όσο θέλει και τα επιβατικά να, τα επιβατικά να ε, υφίστανται περισσότερους περιορισμούς. Κάτι τέτοιο δεν εντάσσεται ε, στην ε, λογική των όσων έτσι με πολύ ανεμικό τρόπο αποφασίστηκαν στην Κομιχάγη. Ε, όταν μιλάμε 100, για 100, στόχο δηλαδή 125 έως το 2020 πρόκειται για ε, έναν στόχο ο οποίος είναι σωστός και δίνει το κατάλληλο κίνητρο γιατί αλλιώς δεν θα συμβαίνει ε, τίποτα δηλαδή θα λένε μια ζωή αυτοκινητομηχανίες όσο μας επιτρέπουν οι νομοθέτες να χρησιμοποιούμε τα παλιά οχήματα αυτό θα κάνουμε δίνουμε εμεί κάποια κίνητρα, κάποιε οθήσει καινοτομία. Εάν δεν δώσουμε αυτά τα κίνητρα, δεν θα υπάρξει καινοτομία. Δηλαδή πραγματικά εγώ εκπλήσωμαι λίγο μετά όσα Mrs. Wills Wills από τους Πρασίνους. Ναι, συγγνώμη, από την ΚΟΕ, από την GUI, συγγνώμη. Ε, και εγώ ε, διαφωνώ με τον κύριο Λαζάκ. Οι εκπομπέ των Ευρωπαϊκών των μεταφορών έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 1999 στο 2007 κατά 26% ενώ η αντίστοιχη μείωση σε άλλους τομείς ήταν της τάξης του 1%. Άρα λοιπόν έχουμε 200 ε, γραμμάδια διοξιδίου του άνθρακα εκπομπέ ε, ανά χιλιόμετρο κατά μέσο όρο αυτή τη στιγμή από αυτή την κατηγορία και κατά συνέπεια κάτι θα πρέπει να γίνει εδώ. Θα πρέπει να δώσουμε σαφή ε, σημάδια εδώ και θεωρώ πως αυτός ο στόχος είναι σωστός όπως τον είχαμε προβλέψει γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε επιτύχει μια μείωση των σχετικών υποπών σε αυτή την κατηγορία ε, κατά 38% πράγμα που αντιστοιχεί με αυτό που επιθυμούμε. Ε, σε ό,τι αφορά την επίτευξη αυτών των 125 ε, γραμμαρίων στο 2020 είναι κάτι τέτοιο το οποίο μπορεί ήδη με την ήδη δηλαδή χρησιμοποιούμενη τεχνολογία να επιτευχθεί. Αυτό είχε αναφερθεί και από την πλευρά ενός εκπροσώπου στην, ε, σε συζήτηση που είχε γίνει και ήδη με κάποιες με κάποια μοντέλα που χρησιμοποιούνται τώρα είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει απλά δηλαδή να γίνουν κάποιε μετατροπέ, κάποιε προσαρμογέ των ε, σημερινών οχημάτων. Άρα λοιπόν το να παρεκκλίνουμε από αυτόν τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2020 δεν τίθεται καν ω ζήτημα. Ω Κοινοβούλιο και ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη νομοθεσία. Στα επιβατικά είδαμε ε, πω η αυτοκινητομηχανία γενικά δεν επιθυμεί αυτή τα να προβεί σε σημαντική μείωση των ασιατικών ε, εκπομπών. Και αυτό ε, μάλιστα μετά από ε, έτη ολόκληρα αλλεπάλληλων δηλώσεων ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο μόνο στους αυτές αυτοκινητομηχανίες. Εάν θεωρούνται πως αυτές οι διατάξεις είναι υπερβολικά αυστηρές, ας υπενθυμίσουμε εδώ πως έχουμε ήδη μειώσει πάρα πολύ τις δικέ μας απαιτήσει. Δηλαδή το, στόχο στόχος των 175 γραμμαρίων έχει μετατεθεί από το 2012 στο 2016. Γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ε, η διαδικασία αν θέλετε τη μείωση τη σχετική ε, ρήπανση. Ε, δεν γνωρίζουμε γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Γερμανία και άλλοι προσπαθούν να αλλάξουν εδώ κάποιου άλλου κανόνε του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά το super credits ε, για να υπάρξει μια τεχνητή, τεχνητή αν θέλετε, μείωση των, της ε, ρήπανσης. Αναφέρθηκαν εδώ και κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά τα αντιχήματα και ούτω καθεξής ως επιχειρήματα. Δεν μπορούμε να κάτι, ένα μέτρο δηλαδή διαφορετικό σε ό,τι αφορά την πραγματική μείωση των εκπομπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όταν κάνουμε αναφορά στα ελαφρά επαγγελματικά προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ταχύτητες, ε, ε, ε, σε ό,τι αφορά την, τις εκπομπές, αναμένουμε και διάφορες μελέτες. Σε βάση περιπτώσει πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν ασχολούνται ακριβώς με αυτό στο οποίο εστιάζουμε. Κατά τη δική μου άποψη, το διοξείδιο του άνθρωπου και βάσει τη δική μου εμπειρία, θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτηση για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Εάν δηλαδή δεν είμαστε λίγο θαραλέοι σε αυτούς τους τομεί, δεν θα χάσουμε μόνο την ηγετική μα θέση ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή, αλλά και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν ενδεχομένως μέσα στα επόμενα, στις επόμενες δεκαετίες να καταστούμε ε, κράτη τα οποία θα εισάγουν αυτή τη τεχνολογία για αυτά τα οχήματα από αμυγός οικονομικής ε, πλευράς δεν θα πρέπει να προσανατολιστούμε αποκλειστικά προς όφελος των ε, αυτοκινητοβιομηχανίων. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες επιστημονικές ε, μελέτες οι οποίες κάνουν λόγο για γύρω στα 135 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε καλού μετρήσιμου στόχου, ώστε ε, να, είναι, να αποφευθούν συγχύσεις και στο μέλλον, να ξέρουμε τι ακριβώ θέλουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα στόχο το οποίο ε, θα πρέπει να ελέγξουμε στα επόμενα πέντε χρόνια για να δούμε τι θα συμβεί. Thank you. For the commission, Mr. Ο κύριος Ρόιν εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τον εισηγητή. Ήταν ευκρινέστατα αυτά τα οποία μας είπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στη θέση της. Νομίζω ότι κανείς σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελε να αφίσταται από αυτό. Τα 175 γραμμάρια είναι νομίζω ένας εφικτός στόχος. Οι αναλύσεις που κάναμε πιστεύουν ότι θα, μας θα οδηγηθούμε εύκολα στα 130 το 2020. Και φιλόδοξο αλλά και εφικτό. Το 135 είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, δύσκολο να το πετύχει κανείς, αλλά δεν είναι κάτι το ανέφικτο. Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα, το θέμα της ε, κατανομής των εισοδημάτων. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύς εκτός θα έλεγα των αρμοδιοτήτων μας και ίσως εκεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών να είχε να πει περισσότερα. Τα λεγόμενα super credits είναι απαραίτητα, είναι ένα κίνητρο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάσταση των οχημάτων από ηλεκτροκίνητα και υβριδικά. Τέτοιου είδους οχήματα θα έχουν σαφέστατο ρόλο να παίξουν όχι ίσω αύριο αλλά μεσοπρόθεσμα. Νομίζω ότι θα υπάρξουν δυνατότητες οι οποίες θα εμφανιστούν σε τομείς όπως ε, το ταχυδρομείο ή και οι παραδόσεις ε, υλικού και προϊόντων σε επίπεδο αστικό. Τα υπόλοιπα θέματα είναι η αλλαγή των ποσοστών για τις εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσει υπάρχουν έτσι και αλλιώ στον κανονισμό για την παραγωγή των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Για μια ακόμη φορά πιστεύουμε ότι ο αριθμός 22.000 είναι ο σωστός. Τα ταχύμετρα και οι περιοριστές ταχύτητας έχει επανέλθει σαν θέμα προσυζήτηση. Έχω δει μια έκθεση η οποία έχει διατυπωθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Πράγματι μειώνει την εκπομπή καυσαερίων και βοηθά και υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει πράγματι ένας έλογος περιορισμός της ταχύτητας, χρήσιμο θα ήταν στα πλαίσια της πολιτικής μας στον τομέα γιατί θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών. Συμπερασματικά είναι σημαντικό το θέμα που έχουμε μπροστά μας νομοθετικά. Οι οδικές μεταφορές αυξάνονται. Ο τομέας ο εμπορικός, ο τομέας των παραδόσεων ε, θα έλεγα είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται σαν δραστηριότητα στο μέλλον και είναι απαραίτητο να το ελέγξουμε το κομμάτι αυτό της κυκλοφορίας και να μειώσουμε τις εκπομπές ε, το 2020 και να έχουμε και ένα μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των εκπομπών από το 2020 μέχρι το 2050 για να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έθεσε πέρυσι τον Οκτώβριο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η στα θα κλείσει τη συζήτηση Βλάσσακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και συμφωνώ με πολλούς από τους ομιλητές. Θα πρέπει οι στόχοι τους οποίους έχουμε να είναι μετρήσιμοι στόχοι. Νομίζω ότι δεν είναι προκλητική η πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά μια πρόκληση βέβαια και εμείς σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προτάσεις αυτές και να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις. Δεν θα πρέπει εμείς να υποκύψουμε αυτόματα στην πίεση την οποία ασκούν οι κατασκευαστές. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η παραγωγή, η παραγωγή καυσαερίων αυτής της κατηγορίας των αυτοκινήτων αφορά το 12% του συνόλου των οχημάτων που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν. Δεν είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά είναι ένα θετικό βήμα. Σχετικά με τους αριθμούς που ακούσαμε, γύρω από την παραγωγή και την κυκλοφορία αυτών των αυτοκινήτων, έχω κάποια στοιχεία από τις αρμόδιες ενώσεις παραγωγών, το 2007 κατασκευάστηκαν 60.000 περίπου και το 2006 συνολικά υπήρχε ένα εκατομμύριο λιγότερο ε, σε επίπεδο αριθμού αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν συνολικά. Ε, τώρα για τον περιορισμό της ταχύτητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή γιατί και μειώνει την εκπομπή Περισσότεροι από εσά είναι οδηγοί, γνωρίζουν ακριβώς και γνωρίζουν ότι μερικές φορές οδηγεί κανείς οδηγεί με 100 χιλιόμετρα και τον προσπερνά ένα τέτοιο ελαφρύ εμπορικό αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό είναι ε, κάτι το επικίνδυνο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε. Δεν έχω άλλα σχόλια να κάνω. Η παρουσίαση, μάλλον το σεμινάριο αυτό στο οποίο αναφέρθηκα, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο, όπως σας είπα, και περιμένω τα σχόλιά σας γραπτά πλέον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνολική ε, λύση. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Μία πολύ απλή ερώτηση θα ήθελα να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά την ε, μείωση τη εκπομπή των σωματιδίων διοξιδίου του άνθρακα. Κοινοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα τομέα των φορτηγών πως η προδιαγραφή Euro 6 σε ό,τι αφορά τα σωματίδια είναι πολύ καλύτερη, δηλαδή προβλέπει μικρότερες εκπομπές, αλλά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου ε, έχει υψηλότερη κατανάλωση από ό,τι προδιαγραφεί Euro 5. Ισχύει αυτό. Αυτό ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα συζητάμε τώρα σε ό,τι αφορά τα ελευθερά επαγγελματικά. Ευχαριστώ. Mr. Rowan. Ο Ρόλε. Υπάρχει μπέρδεμα κάπως με την κατανάλωση Οπότε το Euro 5 και Euro 6 έχουν διαφορετικούς βαθμούς εκπομπών, αλλά όχι του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί είναι μέσα και τα μονοξίδια του αζότου κλπ. Για μένα, Πρόεδρε, ήταν ε, σαφές αυτό. Δηλαδή έχουμε λιγότερο, λιγότερα σωματίδια, υψηλότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Uh, Καλά σας πιστεύω, λέει ο Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Μαΐου. Θα ψηφίσουμε 1η Ιουνίου στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια προβλέπεται να πάει το θέμα τον Ιούλιο. Προς πληροφορία σας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψηφίζει 21 με 23 Ιουνίου. Προθεσμία λοιπόν για κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Μαΐου. Ψηφίζουμε εδώ 1η Ιουνίου όπως σας είπα, στις 21 με 23 Ιουνίου ψηφίζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτό το θέμα και πάει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα στην εμμυρίσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Συνεπώς, Παρακαλώ την καθηγήτρια Σακλίν Μακλέιν να έρθει εδώ παρακαλώ μαζί μας. for the whole debate. Yeah, Okay, colleagues, those who are leaving συνάδελφοι, όσοι αποχωρείτε από την αίθουσα, να αποχωρείτε ησύχως παρακαλώ. Ό,τι πηγαδάκι έχετε, έξω από την αίθουσα παρακαλώ. Θέλω να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Ζακλίν Μαγκλέη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θα μας κάνει την παρουσίασή της και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων μέχρι τις 6 παρατάταρτο, γιατί τότε έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να σας κάνω μια παρουσίαση για την δέκατη επέτειο που έχουμε και που βλέπουμε ότι ο έλεγχος των επιπτώσεων των μεταφορών πάνω στο περιβάλλον είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα και θα σας δείξω μάλιστα ότι μερικές φορές ε, οι εκπομπές ε, των ε, αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί και βλέπουμε και τις απαντήσεις που έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε. Έχουμε 40 δείκτες και βάσει αυτών εξετάζουμε και τι έχει γίνει κατά το παρελθόν για τις εμπορικές μεταφορές, για τις επεμβατικές και σίγουρα θα μπορέσουμε αυτά να τα συζητήσουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες αν χρειάζεται. Τώρα, τι γίνεται σε περίοδο ύφεση. Εννοείται ότι βλέπουμε μειώσεις σε όλους τους τομείς, αλλά ήδη αρχίζουν πάλι <clears throat> να αυξάνονται οι μεταφορές. Τα μηνύματα που υπάρχουν στην έκθεση είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε μαζί. Για τα οχήματα λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι στην έκθεση εντοπίζουμε ότι όταν είμαστε στο 2050-2030 έχουμε όχι μόνο τεχνολογικές βελτιώσεις, αλλά βλέπουμε και τα ωφέλη από τις αλλαγές της μεταφορές και ο συνδυασμός αυτός είναι αναγκαίος. Στα μέτρα για βελτίωση βλέπουμε τεχνολογικές βελτιώσεις στους κινητήρες, στα καύσιμα, στη μείωση των όριων ε, ταχύτητας, πράγμα το οποίο βέβαια συνδυάζονται και με την ασφάλεια. Πάντως, 40-44% μπορούμε να φτάσουμε, κάτι το οποίο δεν φτάνει χρειάζεται ε, μετατροπή των μεταφορών, αλλά χρειάζονται και άλλες δράσεις, όπως περιβαλλοντικές, για παράδειγμα. Όχι μόνο να κοιτάμε τις μεταφορές. Μπορούν λοιπόν να εφαρμοστούν μέτρα, όπως η αλλαγή στις μεταφορές από το ένα είδος στο άλλος, που είναι κλειδί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δίκτυα, σχεδιασμός, διεθνωτικά ταμεία κλπ. Άρα λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την τεχνολογία. Ο συνδυασμό λοιπόν της αλλαγής στον τρόπο μεταφοράς με την χρήση της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και για μείωση των εκπομπών αριών του θερμοκηπίου αλλά και γενικότερα βελτίωση στην κοινωνία και την κινητικότητά της. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τάσεις για συνδυασμό των μεταφορών και με θέματα όπως είναι η χορύπανση. Αλλά βελτιώσεις έχουμε και σε άλλα πράγματα. Όταν κάνουμε υπολογισμούς από το φέλη και τα προβλήματα, αυτά θα τα δείτε στην έκθεσή μας. Υπάρχουν ε, και άλλα ζητήματα. Ε, τα δύο καύσιμα. Η Γερμανία και η Σουηδία έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά τα βιοκαύσιμα, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε τους στόχους μας και να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που δεν θέλουμε είναι να πετύχουμε κάτι σε βάρος άλλων στόχων. Να πετύχουμε ένα στόχο, αλλά καταστρέφοντας άλλους όμως. Πώς επηρεάζει τη χρήση γης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τέτοιοι παράγοντες. Αυτό λοιπόν που πάντα προτείνουμε είναι μια προσεκτική μελέτη επιπτώσεων κάθε φορά για να είμαστε σίγουροι ότι συζητιώνται όλοι οι στόχοι. Και φτάνω και στο τελευταίο που είναι η χορύπανση. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι η χορύπανση και κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Στις πόλεις Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο που ζει εκεί. Άρα δεν πρόκειται μόνο για τις μεταφορές, αλλά πρόκειται και για άλλους παράγοντες που οδηγούν σε ηχορύπανση. Δεν θα ήθελα να δείτε την έκθεση αυτή σαν μια εντελώς αρνητική στάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Πρέπει να προσθέσω ότι σε πολλούς τομείς έχουμε βελτιώσεις, αλλά μόλις έχουμε από μια συζήτηση για το κλίμα, το οποίο τέθη εκεί σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε ότι και άλλα μέρη του κόσμου και η Κίνα και η Ινδία προχωράνε, δεν περιμένουν. Συνδυασμένα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στις πολιτικές μας για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Έτσι πρέπει να δούμε και τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Τρει moment Τρεις ομιλητές, ο κύριος Γκρός πρώτος από το ΕΛΚ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Οι ε, πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε σε στατιστική βάση ε, είναι Λοιπόν, αλλά ε, όπως επανειλημμένα μας λέει ο συνάδελφος Κράμερ, τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω όλα αυτά τα νούμερα. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κάτι. Εδώ μας ε, δίνονται συνέχεια αριθμοί οι οποίοι είναι πάντοτε διαφορετικοί για να ξέρω τι θα συμπεριλάβω στη δική μου έκθεση. Μιλάμε για τις συναλλικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα το 2008. Κάποιοι λένε ότι στη συμμεταφορά ε, από τις μεταφορές προέρχεται το 27% ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι από τις μεταφορές προέρχονται το 24%. ενώ για την ίδια περίοδο ε, θεωρείται το ποσοστό των ε, οδικών μεταφορών ανήκεται στο 80% ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι βρίσκεται στο 70%. Εάν εμεί λοιπόν ως Επιτροπή Μεταφορών βασιζόμαστε σε τέτοιους αριθμούς καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε εσεί ω ανεξάρτητη αρχή ποια είναι τα πραγματικά νούμερα εδώ. Ε, δεύτερη τώρα, πιο άμεση ερώτηση. Όπως διαπιστώσατε και μόλις τώρα από τη συζήτηση που κάναμε, βρισκόμαστε στη φάση α, του πώς α, θα ασχοληθούμε με την τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα. Οπότε θα θέλαμε να γνωρίζουμε ε, α, κατά πόσο οι δικές μας προβλέψεις είναι υπερβολικά αισιόδοξε ή αν πράγματι η τεχνολογία δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Θα θέλαμε να ξέρουμε αυτά που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν για τα φορτηγά και τα οποία συζητήσαμε και για τα επιβατικά αποτελούν κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει, θα μπορούσε να αποτελέσει ρεαλιστικές αξιώσεις, πραγματιστικές αξιώσεις είναι κάτι σχέση με το οποίο πάμε πραγματικά πολύ μακριά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Δεν την έχω διαβάσει με όλες τις, τις λεπτομέρειες, αλλά σας ευχαριστώ που μας την παρουσιάσατε. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και χρόνια βέβαια, που είναι ότι οι μεταφορές ε, είναι υπεύθυνε για ένα μεγάλο βαθμό των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι γνωστό. Οι μεταφορές αυξάνονται επίσης, οπότε η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι πώς μπορούμε με βιώσιμο τρόπο να συνδυάσουμε τις ε, μεταφορές αγαθών και επιβατών με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σαφές ότι για να το καταφέρουμε αυτό χρειάζονται μια σειρά μέτρων, δεν υπάρχει καμία λύση μαγική και γι' αυτό και χρειάζεται η συζήτηση αυτή που κάνουμε φέτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνδυασμό με την πράσινη βίβλο που θα έχουμε αργότερα. Τι μέτρα λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τι μέτρα, περιορισμός ταχύτητας για τα επαγγελματικά οχήματα, να ξέρουμε να επενδύουμε καλά εκεί που έχει νόημα, πώς θα χειριστούμε το εξωτερικό κόστος, να συμπεριληφθεί στον προπολογισμό. Η γνώμη σας ποια είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προτερότητες πρέπει να θέσει για να τις εκτελέσει σε συνδυασμό με τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό πρέπει να ξέρουμε, ποια είναι τα μέτρα τα πιο αποτελεσματικά για να συνδυάσουμε την μεταφορά αγαθών, ανθρώπων με την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μάισνερ από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ε, Καθηγητρία, θα θέλαμε και εμεί από την πλευρά τη δική μα πολιτική ομάδα να σα ευχαριστήσουμε. Δεν είχαμε τη, δυνατότητα ακόμα ε, να διαβάσουμε στο σύνολο τη σχετική έκθεση, αλλά όπω αναφέρθηκε ήδη από του ε, συναδέλφου, θα ασχοληθούμε στο μέλλον πάρα πολύ με το ζήτημα του πώ μπορούμε να μειώσουμε τι εκπομπέ. Ε, και αυτό όχι μόνο μέσω διαφορετικών τεχνολογιών ε, στους ε, κινητήρες όπως κάνουμε στο παρελθόν, αλλά και με άλλους τρόπους. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η μεταφορά των αγαθών θα αυξηθεί μόλις ξεπεραστεί η κρίση και το ζητούμενο εδώ είναι να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους για την υλοποίηση αυτής της μεταφοράς. Ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο υπόψη άλλους, άλλους οδούς μεταφοράς. Για παράδειγμα, η οι ναυτιλιακές μεταφορές ε, είναι κάτι το επιθυμητό. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνούν πάντα όλοι μαζί μας, αλλά ε, για μας δεν είναι πάντα το ζητούμενο να εστιάζουμε στις οδικές μεταφορές. Ε, όμως υπάρχουν ε, κάποιοι Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επίσης σε ό,τι αφορά μεγαλύτερα φορτηγά. Μεγαλύτερα φορτηγά, τα, μεγαλύτερου δηλαδή μήκους τα οποία οδηγούν σε ε, μεγαλύτερη σε, ε, σε μικρότερο αριθμό φορτηγών τα οποία βρίσκονται στους δρόμους. Ε, Επίτρεψέ μου σε παρακαλώ να ολοκληρώσω την παρέμβαση μου. Θα έχεις δυνατότητα να μιλήσω αναφέρθηκε μόλις τώρα πως ε, καλό θα είναι να λαμβάνεται υπόψη η υγεία ε, των ε, ανθρώπων που διαμένουν σε πόλεις και ότι εκεί θα πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία. Στις πόλεις λοιπόν θεωρώ πως υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για τη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων σε σύγκριση με την κίνηση όπως τη βιώνουμε σήμερα η οποία εκπέμπει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν να ληφθούν μια σειρά από μέτρα. Οπότε θα ήθελα να ξέρω να μας πείτε εσείς δηλαδή κατά πόσο θεωρείτε πως θα είχε νόημα το να ξεφύγουμε δηλαδή από τις οδικές μεταφορές και να πάμε προς άλλες, άλλους τρόπους ε, μεταφοράς. ευχαριστώ και ευχαριστούμε και για τα στατιστικά δεδομένα, τα λεπτομερή στατιστικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση δεδομένων, εάν, εάν τα διάβαζαν αυτά τα δεδομένα οι συνάδελφοι εδώ μέσα στην ε, Επιτροπή. Χαίρομαι επίσης ε, πολύ ε, για το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τον όρο αποφυγή, αποτροπή πολύ ενεργά. Γιατί υπάρχουν διαφορές. Αναφέρεται για παράδειγμα η αύξηση των μεταφορών της κυκλοφορίας γενικά ως δείκτης αν θέλετε της οικονομική ανάπτυξη. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει και σε μερικέ ε, περιπτώσει αποτελεί το αντίθετο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιάζουμε στο σωστό στοιχείο. Δεν θέλουμε μόνο μεγαλύτερη ε, απόδοση ε, συνοδευόμενη από όλο ένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα θέλουμε να αποτρέψουμε, να αποφύγουμε ορισμένες συνέπειες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα όσα αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά αυτό το σύννεφο από το ηφαίστειο. Ε, νομίζω πως μας έδειξε ε, το τι ε, συμβαίνει με τις αεροπορικές μεταφορές. Το να έχουμε δηλαδή εισαγωγέ φασολιών από την Κένια, ένα είδος δηλαδή το οποίο καλλιεργείται και στην Ευρώπη, πραγματικά αναρωτιόμαστε. μήπως ε, ε, η κατάσταση εδώ είναι λίγο ε, στριβλωμένη. Το ότι δηλαδή είδαμε να μην υπάρχουν κάποιες προμήθειες ορισμένα αγαθά μας ε, δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει μία πτυχή της ανάπτυξης η οποία πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε κατά πόσο έχει νόημα και την οποία εγώ καταδικάζω ως οικολόγος ε, και η οποία θα πρέπει να αμφισβητηθεί γενικότερα σε σχέση με τις ε, φορολογικές διευκολύνσεις οι οποίες παρέχονται στον αεροπορικό τομέα. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι θεωρείτε σε σχέση με την άποψη της Ροζίνης. ή μάλλον ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρήση αυτού του καυσίμου ε, θεωρείτε δηλαδή πως έχει νόημα να προωθούμε τέτοιου είδους μεταφορές υπό αυτούς τους όρους. Ένα ε, ακόμα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την κυκλοφορία αφορά και το ζήτημα του θορύβου από, τις, από την κυκλοφορία. Είδαμε δηλαδή ότι κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι διέμεναν κοντά σε αεροδρόμια άκουσαν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό πουλιά και πάλι να τελαϊδούν. Ε, μάλλον αυτό δεν θα το βιώσουν ε, πλέον ε, σύντομα στο εγγύς μέλλον. Τι συμβαίνει για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον θόρυβο από αεροπλάνα. Ε, ήδη υπάρχουν κάποιες ε, κλήσεις από την πλευρά ε, των Ηνωμένων Πολιτειών να μειώσουμε αν θέλετε λιγότερο, λίγο παραπάνω τις απαιτήσει που έχουμε απέναντι σε αεροπλάνα αμερικανικά σε ό,τι αφορά το θόρυβο. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Θέλετε να προσπαθήσετε να δώσετε απαντήσεις στην πρώτη σειρά των ερωτήσεων και θα ακολουθήσει και δεύτερη. Οι αριθμοί που έχετε μπροστά σας αφορούν το 2007. Νομίζω ότι είναι αρκετά κατάλληλη για την τεκμηρίωση των πολιτικών τους οποίους ακολουθούμε. παρατηρείτε όμως επίσης ότι στην αρχή της παρουσίασης περιλαμβάνουμε και κάποιους αριθμούς που δείχνουν ότι μπαίνουμε σε ύφαση Είναι αριθμοί βέβαια οι οποίοι απλά ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν κάπως σχετικοί δείκτες. Έχουμε εξυπηρετήσει το 90% των υποχρεών μας σε σχέση ε, με το Κιώτο από το 2008 και 2009 θα δείτε ότι μειώνεται η συμμετοχή κάποιων μορφών μεταφορών και από κάποια στιγμή και μετά αυξάνεται όμως πάλι. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και από πηγές των Ηνωμένων Εθνών κάποια τα οποία να είναι σχετικά αξιόπιστα. Νομίζω επίσης ότι αν αναφερόμαστε σε 70 ή 80% δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι σαφές ότι των, το ποσοστό των οδικών μεταφορών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για τις ε, τελευταίες ερωτήσεις. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον όγκο, στις αλλαγές της ενέργειας, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε. Υπάρχουν πολύ λίγα μεμονωμένα μέσα τα οποία δίνουν κάποια στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα. Ένα από αυτά τα οποία εξετάζουμε είναι οι επιδοτήσεις. Αργά ή γρήγορα οι επιδοτήσεις σχετικές δηλαδή με φόρους γύρω από τα καύσιμα θα πρέπει να συζητηθούν. Είναι ενδιαφέρον όταν βλέπει κανείς τις εσωτερικές ε, μεταφορές παραποτάμιες και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες οι οποίες δεν έχουν ακόμα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Από την άλλη όμως, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα αυτά περισσότερο, απαιτούνται πάρα πολλές επενδύσεις για να υπάρξουν γρήγορες λύσεις. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν οι βιομηχανίες μας να προτείνουν νέες τεχνολογίες. Αν δείτε όμως κάποιες από τις καμπύλες στην έκθεση, βλέπετε ότι οι βελτιώσεις αυτές προέρχονται και από βελτιωμένη σχεδίαση των μηχανών, αλλά πάντα ε, ζητάμε στα μέσα του 21ου αιώνα να έχουμε φτάσει στο 90% στη μείωση των καυσαερίων. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε λάβει δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν εκ νέου τον ρόλο των περιφερειακών ταμείων και δεν θα πρέπει να περιμένουμε τα αποφάσεις των άλλων, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε εξ αρχής να επηρεάσουμε ε, μια πολιτική η οποία να χαρακτηρίζεται από συνοχή, να λύσουμε προβλήματα όπως το καμποτάζ και ταυτόχρονα να βρούμε τις πιστώσεις για, τα, για τους ιεροδρόμους υψηλής ταχύτητας που όλοι ξαφνικά ξανααγαπήσαμε τις τελευταίες εβδομάδες με τα προβλήματα στις αερομεταφορές. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, το κόστος τότε θα είναι κάποια στιγμή ιδιαίτερα υψηλό. Σε επίπεδο περιβάλλοντος πόλεων Υπάρχουν άμεσα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, πολεοδομικά, διόδια, απαλλαγή από φόρους για ηλεκτροκίνητα οχήματα και οι δυνατότητες βέβαια για επενδύσεις εδώ μας διαφεύγουν. Η Ευρώπη ε, συνεργάζεται, ξέρετε, υπεγράφει μια συμφωνία με την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Cherry για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αυτά είναι τα αυτοκίνητα που θα δούμε ε, στις δικές μας χώρες. Τι θα είναι, Κινέζικα, Πεζό ή κάτι άλλο. Υπάρχει επίσης ε, ένα νορβηγικό αυτοκίνητο το οποίο κατασκευάζεται στη Φιλανδία και νομίζω ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά είναι οικολογικό, ιδιαίτερα ελαφρύ, μικρό, χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένα υλικά και έχει ανοίγει νέες προοπτικές. Τα ρεύα. Δεν είμαστε κατά των μεταφορών, ίσα ίσα η κινητικότητα είναι αυτό το οποίο θέλουμε να εγγυηθούμε, αλλά θέλουμε να εγγυηθούμε τη σωστή μορφή, προστατεύοντας το περιβάλλον από μόλυνση και από ε, θορύβους. Νομίζω ότι ε, είμαστε σύμμαχοι στους στόχους τους οποίους έχετε και έχουμε. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό περιβαλλοντικό επίπεδο και στις πόλεις μας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις από τη μόλυνση και την ηχητική μόλυνση επίσης. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας προς την κατεύθυνση αυτή, έστω και σε αυτή τη φάση. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι μετά από τη συζήτηση για τα ελεύθερα ε, επαγγελματικά και, τις, ε, και τους αντίστοιχους ε, περιορισμούς για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα να δίνουμε την ευκαιρία τώρα στον επιστημονικό τομέα να εκφράσει τη δική του άποψη. Ε, και γνωρίζουμε πως ε, ε, όταν έχουμε τέτοιου είδους καύση προφανώς και θα προκύπτουν θα προκύπτουν και εκπομπές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργούμε ε, προσδοκίες. Και αν λέμε ότι έχουν φτάσει οι κινητήρες στο επίπεδο που μέσα, μέχρι το 2050 θα, έχουμε, θα επιτύχουμε περαιτέρω μείωση κατά 9% και όχι παραπάνω, ε, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει. Δηλαδή όλα αυτά σχετίζονται, εκπομπές δηλαδή και με τις, ε, ε με τις ε, διακοπές, η ίδια η η αναζήτηση ενός χώρου στάθμευσης, μια θέση στάθμευσης ε, ε, αποτελεί την αιτία για το 20% ε, των εκπομπών σε ό,τι αφορά τις πόλεις, δηλαδή και οι τρόποι ζωής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές εκτιμήσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, των e-cars, ε, όχι μόνο για τον, ε, για τους, ε, αστικό τομέα. Η χρήση μπαταριών λιθίου είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα και η απόδοση ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι πολύ κακή, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, χρειάζομαι μια τεράστια μπαταρία για να μπορέσω εγώ ίδιος να μετακινηθώ χωρίς να έχω επιβάτες πάνω στο, όχημα. Ε, εγώ ε, σκέφτομαι εδώ ότι θα, ότι πρόκειται εδώ για μια μεταβατική λύση που αυτή θα αντικατασταθεί από, την, από νέα μονάδα καύσης. η οποία πλέον δηλαδή με υδροκίνητα αυτοκίνητα θα οδηγήσει στο να έχουμε καύση νερού που σημαίνει καμία εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Ε, επίσης και σε σχέση με τα ε, γνωρίζω πως προσπαθούμε να επιτύχουμε τέτοιου είδους ε, οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα, ε, για τα οποία δεν θα χρειάζεται αυτά να επαναφορτίζονται σε συγκεκριμένου ε, χώρου, σε συγκεκριμένα πρατήρια, αλλά να υπάρχει κατά μήκο των αυτοκινητοδρόμων μια τροφοδοσία. Ευχαριστώ. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ καθυστέρησα λίγο. Αλλά να ξέρετε ότι έτσι αλλιώς παρακολουθούμε τις εκθέσεις του οργανισμού σας με ιδιαίτερη προσοχή. Έχω μερικές ερωτήσεις. Από τα διάφορα μέσα, που βέβαια δυσκολευόμαστε εμεί με την επικουρικότητα να εφαρμόσουμε τα σχέδια, εν πάση θέλω να ξέρω κατά πόσο ο οργανισμός αν περιλαμβάνει και το θέμα των αποστάσεων. όχι τόσο για τις επιβατικές όσο για τις εμπορικές, την απόσταση ανάμεσα στην περιφέρεια και το κέντρο. Είναι αυτό ένα κριτήριο, πιστεύουμε εμείς, σημαντικό που χρειάζεται να μελετηθεί περισσότερο επιστημονικά στη Γαλλία. Ας πούμε, ξέρω ότι υπάρχει ένα μοντέλο <clears throat> για να υπολογιστεί η απόσταση αυτή της περιφέρειας από το κέντρο. Και θα ήταν ενδιαφέρον ότι έχουμε και για την Ευρώπη, μάλιστα τη διευρυμένη Ευρώπη, για τις πόλεις τώρα, τον αστικό χώρο. Θέλω να ξέρω, ο οργανισμός θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο. Τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν να πάρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα τι θα χρησιμοποιήσουν ε, μετρό, ε, τραμ, Μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε για το τι είναι καλύτερο και τι όχι. Τέλος, πράσινη απασχόληση. Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βελτιώνοντας τα κριτήρια τάσεων. Να ξέρουμε δηλαδή και για τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Τέλος, βλέπω και κάτι όσον αφορά τα όρια ταχύτητος. Περιορισμός των εκπομπών, εφόσον περιοριστεί η ταχύτητα, και ασφάλεια στους δρόμους, βέβαια. Στην Βαρκελόνη όμως θυμάμαι ότι όταν βάλαμε τα 80 χιλιόμετρα την ώρα στον χώρο γύρω από την πόλη, τελικά δεν διαπιστώσαμε μείωση των εκπομπών. Μπορεί να οφείλεται σε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Υπάρχουν ε, ε, μοντέλα αξιόπιστα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι η εκπομπή των ε, οχημάτων ή πως και η χρήση που γίνεται στα Όσο περισσότερους στόχους βάζουμε για τη μείωση των ε, οχημάτων, από την άλλη αυξάνουμε τον αριθμό των χιλιόμετρων που διανύονται και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να ταυτίσουμε τους δύο στόχους αυτούς, μείωση των εκπομπών στη στιγμή της παραγωγής, αλλά από την άλλη και μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων γιατί συνεχώς αυξάνονται ε, τα χιλιόμετρα που διανύουν. Τώρα, σχετικά με τους λεγόμενους κύκλους πόλεων. Πράγματι μπορεί και μέσω της πολεοδομίας, η οποία δεν είναι, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, να βρεθούν κάποιες λύσεις. Τι θα γίνει με τα λεγόμενα, όχι μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα τα οποία είναι κοινή χρήσεω να μην υπάρχει δηλαδή ατομική ιδιοκτησία οχημάτων, αλλά να υπάρχουν δυνατότητες χρήσης αυτοκινήτων, γιατί μέσα στις πόλεις, τις μεγάλες, δεν υπάρχει δυνατότητα απέρετσέρο παρουσίας πολλών αυτοκινήτων. Κάθε οικογένεια έχει ένα, δύο και τρία αυτοκίνητα. Είναι ανυπόφορο αυτό, ιδιαίτερα σε σχέση με την λεγόμενη κατανομή του χώρου των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητα μεν, αλλά τα αυτοκίνητα που μοιραζόμαστε με άλλους. Ένα αυτοκίνητο δηλαδή, ένα όχημα που είναι στη διάθεσή μας, που επιτρέπει στον πολίτη της πόλης να μετακινείται είτε με τα μέσα ε, κοινή μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, είτε με τραμ, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, αλλά να χρησιμοποιεί φυσικά και ε, τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμεύουν σε πολλούς χρήστες κάθε φορά. κύριος Καντσιάν. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα πρέπει να βασίζεται σε δύο ε, βασικές έννοιες. Από τη μία η διαλειτουργικότητα και από την άλλη ε, το επιμελητιακό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε μια επιμελητία η οποία να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην οργάνωση και στον εξορθολογισμό των μεταφορών. Αν το πετύχουμε αυτό θα έχουμε κάνει ένα βήμα αρκετά σημαντικό προς τα εμπρός. Να σας μεταφέρω τις εμπειρίες που έχουμε από το Ιντερπόρτο της Πάντοβα, όπου έρχονται εμπορεύματα από το κέντρο της Ιταλίας και προς, προς το κέντρο της πόλης μάλλον ε, φεύγουν ε, τα προϊόντα αυτά μόνο με ηλεκτρικά μέσα. Αυτό έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα στην πόλη της Πάντοβα είναι κάτι το οποίο είναι τμήμα αυτών των περίπλοκων κανόνων, εν πάση περιπτώσει, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Το λογισμικό θα πρέπει να ακολουθεί και αυτό έτσι ώστε οι μεταφορές να γίνονται από οχήματα τα οποία να είναι γεμάτα και όχι άδεια. Όταν παρουσιάστηκε η τελευταία προεδρία, ε, βασικός στόχος ήταν, θα έλεγα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το θέμα είναι σημαντικό, θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να το βάλουμε στις ρωμαϊκές καλένδες, όπως είχαμε κάνει παλιότερα με το υδρογόνο, αλλά αν για να περάσουμε στο, στο ηλεκτρικό πλήρως αυτοκίνητο πρέπει να περάσουμε από το υβριδικό, αυτός είναι ένας δρόμος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να διανύσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ, θέλετε ξανά να πάρετε το λόγο. Ναι, λέει κυρία Μάισνερ. Ναι, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με ένα τομέα τον οποίο δεν θίξαμε ακόμα. Ήδη αναφερθήκαμε σε άλλα, άλλους ε, τρόπους ε, μεταφορών ή ε, δεν ξέρω άλλους κινητήρες αλλά ιδιοχημάτων οχημάτων και ούτω καθεξής αλλά από τις κυκλοφορικές συμφορήσεις δημιουργούνται όχι μόνο εκπομπές αλλά και θόρυβος. Ίσως καλύτερα συστήματα κυκλοφορία θα μα βοηθούσαν τόσο να επιτύχουμε μείωση αυτού του θορύβου, Ασχέτω ε, δηλαδή των εκπομπών και ασχέτω ε, του αριθμού των οχημάτων. Ε, πώς θεωρείτε πω θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε εδώ τι επιδόσεις μα. Ευχαριστώ για την υπομονή σα, Πρόεδρε. Εγώ μίλησα για το τραμ γιατί μου φάνηκε πιο τίγωνα, αλλά δίκαιο έχει και ο συνάδελφο. Λοιπόν, κυρία Μαγκλίν. Τι δυνατότητες υπάρχουν να μας βοηθήσει ο οργανισμός, και αναφερθήκατε σε αυτό, στον έχουμε ένα δεύτερο κύκλωμα κινητικότητας στην περίπτωση που, να, κλείνουν τα αεροδρόμια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος κάποια στιγμή όπως αυτές τις 4-5 μέρες που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισαν οι ευρωπαϊκοί εθέρες, μήπω θα μπορούσε να γίνει κάποια μελέτη ή κάτι να βάλετε στην επόμενη έκθεσή σας για να δούμε πώς και εμείς θα μπορούσαμε να βάλουμε σαν σύσταση να υπάρχει ένα δεύτερο κύκλωμα κυκλοφορίας με τρένα ή να μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε αποστάσεις τις οποίες συνήθως διανύουμε με αεροπλάνα, με τα τρένα για παράδειγμα υψηλών ταχυτήτων, κάτι τέτοιο. Πριν απαντήσετε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι χθες μπήκα σε ένα υβριδικό αυτοκίνητο που δούλευε με ηλεκτρισμό αλλά όταν τέλειωσε η μπαταρία πήρε μπρος η μηχανή, γέμισε την μπαταρία και μετά ξαναπήρε μπρος η μπαταρία και νομίζω ότι αυτό λύνει τα προβλήματα που έχουμε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία μετά από 25 λεπτά λειτουργίας χάνουν την ε, ηλεκτρική ενέργεια. Ένα άλλο σημείο το οποίο ήδη νομίζω στο οποίο αναφερθήκατε είναι ότι την τελευταία εβδομάδα τα τρένα υψηλής ταχύτητας φάνηκαν όλα ιδιαίτερα ελκυστικά γιατί δεν υπήρχαν αεροπλάνα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω σαν κάποιος ο οποίος τα, τα Χριστούγεννα με έστησαν τα τρένα υψηλής ταχύτητας ότι τα αεροπλάνα ήταν πάρα πολύ ελκυστικά και μας ωφέλησαν πολύ. Απλά ήθελα να το σημειώσω. Ε, του σε πρόεδρε, του σε. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Όπως είπα και εγώ προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα της διασφάλισης της κινητικότητας και της μείωσης των εκπομπών και λύνοντας μάλιστα και άλλα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε κάποιες σοβαρές και δύσκολες επιλογές. Κατανοώ το θέμα της επικουρικότητας, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει το ρόλο της. Πού ακριβώς είναι τα κέντρα παραγωγής, πού θα πρέπει να έρχεται το εμπόρευμα, προς τα πού θα πρέπει να πηγαίνει, να συγκεντρώνεται και να στηρίζεται. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά που βλέπει κανείς όταν συζητά τα θέματα του κλίματος κτλ είναι ότι όλες οι περιοχές της Ευρώπης δεν θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα κέντρα παραγωγής, αλλά κάθε περιοχή θα έχει τη δική της οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα τον προγραμματισμό των μετακινήσεων, ιδιαίτερα ε, τα εμπορεύματα και την επιμελητία που τα συνοδεύει. Νομίζω ότι αυτό είδαμε και σε άλλους τομείς. Όταν κάνει κανείς τα μέσα, τους μηχανισμούς πιο αποτελεσματικούς, ο καταναλωτής στην ουσία αγοράζει ένα ισχυρότερο μηχανισμό. Δηλαδή όταν κάνουμε κάτι πράσινο, τότε ο καταναλωτής αγοράζει πιο ισχυρά οχήματα ε, και συνεπώς ακυρώνουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χρόνος τον οποίο έχει ο καταναλωτής στη διάθεσή του για να μετακινηθεί και μπορεί να πει ότι εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε και για μία ή μία μισή ώρα την ημέρα για να πάμε στη δουλειά μας, μπορούμε να μένουμε και πολύ μακριά από τις πόλεις μέσα σε ωραία τοπία. Υπάρχει λοιπόν και αρνητική πλευρά όταν κάποιος προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα πιο αποδοτικά για τις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στα πλαίσια ε, της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας σήμερα παράγονται οχήματα τα οποία είναι κάτω του 100. Βέβαια δεν έχω δει μέχρι τώρα καμία ηλεκτρική Φεράρι και εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα την αγοράσω όταν κυκλοφορήσει και θα σας πάω βόλτα πρόεδρε άμα την έχω. Υπάρχουν λοιπόν δεν χωράω σε μια Φεράρι λέει ο προεδρό. Πάντως απαιτείται χρόνος, πρέπει να υπάρξουν κάποιε επιδοτήσει για την αγορά. Τα υβριδικά είναι χρήσιμα σαν υποκατάστατα, τα ηλεκτρικά έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν. Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι τόσο, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν. Ναι, μεν οι μπαταρίες βελτιώνονται συνεχώς, Υπάρχουν σε πόλεις ε, όπως η Κοπενχάγη ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν για 4-5 ώρες και θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικά. Ελάτε στην Κοπενχάγη να τα δείτε. Νομίζω πάντως ότι σε όλους τους τομείς, τους κινητήρες, τις μπαταρίες, τα υβριδικά, στα ηλεκτρικά, όλοι οι τομείς έχουν τον ρόλο να παίξουν, καλούνται να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, έναν ρόλο καινοτομικό, μέσω και της δημιουργίας ε, των ε, υποδομών. Ε, τα μετρό, τα τραμ, ξέρετε ότι υπάρχουν περιοχές είτε αντισυσμικές κτλ που δεν μπορούμε να φτιάξουμε μετρό. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ελαφρών τραμ σε πάρα πολλές πόλεις με πολύ χαμηλό κόστος, κάτι το οποίο θα μειώσει τις μετακινήσεις με ιδιωτικά αυτοκίνητα σε ημερήσια βάση δεν είμαι εγώ υπέρ ε, του συστήματος των επιδοτήσεων γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν εισαχθούν τα συστήματα αυτά χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποσυρθούν μετά. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορεί κανείς να μην δίνει διαταγές αλλά μπορεί να δίνει κατευθύνσεις για το πού μπορούμε να πάμε. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να δώσουμε κίνητρα για να αλλάξουν οι, οι νοοτροπίες και οι διαδικασίες μετακίνησης Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να φανούμε ε, πιο αποτελεσματικοί για τις πράσινες θέσεις εργασίας και στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα. Αν ε, κανείς ε, βάλει κάποιους αριθμούς που έχουμε στη διάθεσή μας στον τομέα των πράσινων θα έλεγα αυτοκινήτων, θα δείτε ότι στην Κίνα δημιουργούνται πάρα πολλές τέτοιες θέσεις. Έχουν συνδέσει ας πούμε ε, τα ηλεκτρικά ποδήλατα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο το οποίο θα δώσει τεράστιους αριθμούς ποδηλάτων τα οποία φορτώνονται τη νύχτα, φορτίζουν συγγνώμη τη νύχτα για τις δημόσιες υπηρεσίες στην Κίνα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα θέμα στην Ευρώπη, πρέπει να τα ταξινομήσουμε κάπως τα θέματα και τις ευκαιρίες μεταφορών που έχουμε. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες οικονομικές που θα πρέπει και αυτές να τις εκμεταλλευτούμε. Νομίζω ότι η διαλειτουργικότητα και τα επιμελητιακά στοιχεία του συστήματος των μεταφορών. Αν δει κανείς τη Σκανδιναβία βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αποτελεσματικές εταιρείες μεταφορών είναι τόσο σαφή τα ωφέλη που ε, νομίζω ότι αν ξεκινήσει κανείς να δουλεύει προς την κατεύθυνση αυτή δεν απομακρύνεται πλέον μετά. Τώρα για το αν θέλουμε ένα εναρμενισμένο σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Όχι. Αυτό το οποίο όμως χρειαζόμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η υπηρεσία μου είναι κάποιες οδηγίες, κάποιοι χάρτες ε, έτσι ώστε να βλέπουν οι πολίτες ε, τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιούν, ε, πού βρίσκονται τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτή την τεκμηρίωση θα πρέπει να την έχουμε απόλυτα διαθέσιμη για το σύνολο του τομέα των μεταφορών. Παρά τις διαφορές λοιπόν που υπάρχουν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στοιχεία στην διάθεσή μας και συγκεκριμένες προτάσεις ιδιαίτερα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερο. Δεν θα ήθελα άλλη μια κρίση με ε, ηφαιστειακή τέφρα πάνω από τα κεφάλια μας. Όταν ξανασυμβεί ελπίζω να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ε, δυνατότητες που έχουν οι αερομεταφορές έτσι ώστε ε, να μην νιώσει το κοινό την ανασφάλεια την οποία βίωσε. Ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι αν υπάρξει μια νέα τέτοια, ένα τέτοιο φαινόμενο θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα, ε, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι το θέμα και το πώς το παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τις απαντήσεις σας Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 το πρωί. Οι συντονιστές ξεκινούν σε 15 λεπτά.